Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, ας αρχίσουμε τις εργασίες μας. Καταρχήν σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, γιατί προηγήθηκε η συνεδρίαση των συντονιστών, που ήταν απαραίτητη και παρατάθηκε λίγο περισσότερο από το αναμενόμενο, γιατί έπρεπε να εξετάσουμε τι θα γίνει μετά την αποτυχία της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό το 2013. Ήταν από τα βασικά στοιχεία της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε αρκετά φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Θα προσπαθήσουμε να την διεκπαιρεώσουμε ε, προσπαθώντας να εργαστούμε γρήγορα και καλά. Το γοργόν και χάρη έχει, χωρίς βέβαια να περικόψουμε τα σχόλιά μας και χωρίς να στερηθούμε τη δυνατότητα να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Μερικοί συνάδελφοι ζήτησαν να να συζητηθούν νωρίτερα τα σημεία τους, αλλά επειδή έχουμε ήδη μια μικρή καθυστέρηση, να διαφυλάξουμε πρώτα το χρόνο της ψηφοφορίας από τη στιγμή που εξασφαλίσουμε την τήρηση της ώρας ψηφοφορίας μπορούμε να συζητήσουμε λίγο νωρίτερα το σημείο 9 του κυρίου Αλφόνση με την κυρία Καρβάγιο Σκιώδη Συγκεντρία. Ανακοίνωση του Προέδρου. Μία προφορική ανακοίνωση. Υπάρχει, στο... υπάρχει μόνο στο δικό μου κομπονιούς η ανακοίνωση αυτή. Στο δικό σας δεν υπάρχει. Γιατί ο Πρόεδρος έχει μια πληροφορία που εσείς δεν την έχετε ακόμη, αλλιώς δεν θα ήταν Πρόεδρος. Εκ μέρους της κυρίας Σίγκε Γκρέσλε που απουσιάζει γιατί έχει αναλάβει ένα πολύ λεπτό και πολύ σημαντικό άλλο θέμα για την ε, Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και μου ζήτησε να τη αναπληρώσω σήμερα για το θέμα του δημοσιονομικού κανονισμού σε ό,τι αφορά τη κατεξουσιοδότηση πράξη. Θα διαβάσω το κείμενο της στα αγγλικά. Η κατεξουσιοδότηση πράξης ε, έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 29 Οκτωβρίου. Θα, έπρεπε, θα πρέπει να ισχύσουν από την 1η η 2013 μαζί με το δημοσιονομικό κανονισμό. Θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ μόνο εφόσον δεν υποβληθούν στάσεις, είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο μέσα σε ένα δίμηνο από την κοινοποίηση. Για πρώτη φορά οι δύο επιτροπές ελέγχου προπολογισμού και κόντ με βάση το άρθρο 51 έλαβαν από κοινού ε, κατεξουδότηση πράξης για εξέταση. Η κυρία Γκρέσλε παραλαμβάνω ακολύεται για σήμερα, αλλά μου ζήτησε να σας ε, διαβιβάσω τις ε, αφιβολίες της σε ό,τι αφορά την ομιμότητα του άρθρου 21 του RAP, των εφαρμοστικών κανόνων δηλαδή, σε σχέση με τη δημοσίευση των κανόνων των δικαιούχων σε περίπτωση που είναι ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα. Τώρα, στις διαπραγματεύσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρήσω ότι όχι μόνο θα πρέπει να ε, δημοσιευτούν τα ονόματα των δικαιούχων του, τους περιοχής ΝΑΤ2, αλλά και ε, οι επαρχίες ε, Land Landkreis, Arrondissement, County, δηλαδή υποπεριφερειακές ε, ζώνες, ενότητες. Για να διευκρινιστούν τα σημεία αυτά, θα πρέπει να, να συγκαλεστεί μια νέα συνεδρία της ομάδας εργασίας στο Στρασβούργο στις 21 Νοεμβρίου με το θέμα αυτό, όπου ο κύριος Μπουταρέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μπουταρέλη δεν είναι ποδοσφαιριστής Ιταλός. Αχα, όχι, όχι είναι ε, υποδιευθυντής του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων. Θα μας κάνει ενημέρωση για το θέμα αυτό ο Μπουταρέλη. Αν ε, θέλουμε να υποβάλουμε στάσεις αντιρρήσεις, θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε το αργότερο στις 3 Δεκεμβρίου. μαζί με την Επιτροπή Κοντ. Γι' αυτό προτείνω να θεσπίσουμε την διορία για να υποβάλουμε και αιτιολογημένο ψήφισμα, αν θέλουμε να υποβάλουμε έσταση, και να ορίσουμε την προθεσμία αυτή στις 22 Νοεμβρίου. Έχουμε λοιπόν 8 μέρες στη διάθεσή μας. Αυτά ως προς την ενημέρωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διερμηνία. Πριν είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, δεν είχαμε διερμηνία, αλλά στο μεταξύ δεν βλέπω καμία αντιρρήση, αλλά είτε δεν με ακούει κανένας, είτε στο μεταξύ έχει αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα και μπορούμε να συνεχίσουμε. Και λειτουργεί και το web streaming, η αναμετάδοση απευθείας μέσω του, του δικτύου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έγκριση των πρακτικών, θα πρέπει να ε, να εγκρίνουμε και τα πρακτικά της 18ης Οκτωβρίου, ώστε οι ψηφοφορίες για το ΤΑΠ 5 και το Ταμείο Αλληλεγγύης να προσδιορίσουμε ότι ήταν ψηφοφορίες πολιτικού προσανατολισμού και όχι επίσημης έγκριση των δύο κειμένων. Γιατί σήμερα το απόγευμα θα ψηφίσουμε επίσημα τα δύο κείμενα. Προηγουμένως ε, κολλιόμασταν νομικά γιατί δεν ε, είχε αποφαθεί το Συμβούλιο. Πριν από δύο μέρες επισημοποίησε τη θέση του Συμβούλιο, οπότε μπορούμε και εμείς σήμερα επίσημα να ψηφίσουμε. Οπότε, ναι και δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την αλλαγή αυτή, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4 της ημέρησης διάταξης. Τα αποτελέσματα δηλαδή της συνδιαλλαγής και μάλιστα η αποτυχία της συνδιαλλαγής της 9ης Νοεμβρίου. Βέβαια, δεν α, μας εμπόδισε η αποτυχία αυτή να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μέχρι την Τρίτη το βράδυ. Αλλά άκαρπες ήταν και ε, οι παρατεταμένες αυτές τις διαπραγματεύσεις και έτσι διαπιστώσαμε τελικά την αποτυχία της συνδιαλέγησης. Δεν θα επανέλθω στις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η διαπραγμάτευση αυτή, η συνδιαλέγη, γιατί σχεδόν όλοι οι παρόντες παρακολούθησαν το θέμα αυτό ένεργα και ήταν και μέλη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή της Συνδιαλέγης. Άρα γνωρίζετε όλοι από ό,τι περάσαμε και Ακούσατε και τις δηλώσεις, μερικοί μάλιστα υποβάλλατε και εσείς πολιτικές δηλώσεις που κρίνατε σκόπιμο να κάνετε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας, αλλά να κάνω πρώτα μια σύντομη παρουσίαση. Ποιες είναι οι μελλοντικές μας προοπτικές. Αυτή τη στιγμή δεν κατέστη δυνατό να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπει η συνθήκη για την υιοθέτηση, για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2013 εξαιτία ε, ενός πολιτικού αδιεξόδου που δημιουργήθηκε για τον τρόπο πληρωμής ε, των εξόδων που θα πρέπει να γίνουν ή που σε μεγάλο βαθμό έγιναν ήδη και θα πρέπει να αποζημιωθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 και πρέπει οι λογαριασμοί αυτοί να πληρωθούν μέχρι το, τα τέλη του 2012 γιατί αφορούν ελλημένες υποχρεώσεις είτε δαπάνες που έχουν ήδη γίνει. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν καθαρή και εξάστερη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμησε ότι πέρυσι όταν, εξετάσαμε το, όταν εγκρίναμε τον προϋπολογισμό του 2012 γνωρίζαμε και μας το είχε επισημάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζαμε ότι αναλαμβάναμε τον κίνδυνο να διαπιστώσουμε στα, μέσα της χρονιάς ότι οι πιστώσεις πληρωμών δεν επαρκούσαν για να, ανταποκριθούν, να, να δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες μας. Και ιδιαίτερα για τα διαρθρωτικά ταμεία και για να ε, πληρωθούν οι λογαριασμοί που έγιναν. Ε, πρόκειται για δαπάνες που έγιναν δηλαδή από τα κράτη-μέλη, από τις εθνικές ή ε, περιφερειακές ε, αρχές των κρατών μέλων. Και άλλωστε ο δημοσιονομικός κανονισμός υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποζημιώσει μέσα σε ένα δίμηνο τα κράτη-μέλη για τις ανηλυμένες δαπάνες. Και για να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος και με πρωτοβουλία του ίδιου του Συμβουλίου, συμπληρώσαμε τη συμφωνία για τα ποσά του προπολογισμού με μια κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων. Αυτή η κοινή δήλωση ήταν σαφέστατη. Αναλαμβάναμε τη δέσμευση σε περίπτωση διαπίστωση έλλειψη των πιστώσεων πληρωμών, να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει πάρα ένα σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού και μάλιστα το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αναλάμβαναν την υποχρέωση να το, να το εξετάσουν το συντομότερο δυνατό. Ήδη από τον Οκτώβριο διαπιστώθηκε σχεδόν πλήρης ε, εξάντληση των, των πιστώσεων πληρωμών για τα πιο σημαντικά κοινοτικά προγράμματα. 8 δισεκατομμύρια, 300 εκατομμύρια για, το, για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, ποσά που έπρεπε να επιστραφούν στα κράτη-μέλη και μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια για προγράμματα που διαχειριζόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και μάλιστα πρέπει να πληρωθούν 45 μέρες μετά την υποβολή του λογαριασμού. Οι δεμή ε, οφείλονται οι περιμερίες. Ιδιαίτερα το lifelong learning, το έρασμό και το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο. Πέρυσι ήταν περίπλοκες οι διαπραγματεύσεις και περιπλάξαν τελευταία στιγμή γιατί τα ποσά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά τις ε, ανάγκες ε, της πιστώσης πληρωμών για το Τέλο του είχαν, δια... είχαν αφισβητηθεί αυτά τα ποσά από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό είπαμε ότι φέτος θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να συμφωνήσουμε εκ των προτέρων για τα πώ θα εκτιμήσουμε τις ανάγκες των πιστώσεων πληρωμών, ώστε να αποφύγουμε ε, περιπλοκές αντίστοιχες και για τον προϋπολογισμό του 2013 τεχνική περιπλοκή δεν ανέκυψε φέτος. Μια πρώτη πρόεδρος, πρόοδος και μας ικανοποίησε ιδιαίτερα αυτό. Βέβαια, βρεθήκαμε ε, μπροστά σε μια απρόπτη κατάσταση, γιατί καμία αντιπροσωπεία και το είχα διευκρινίσει δύο φορές στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής και στις 27 χώρες μέρες, καμία αντιπροσωπεία φέτος δεν αφισβήτησε δημόσια και επίσημα και για τα δημοσιονομικά θέματα όλα είναι ανοιχτά και φανερά και δημόσια. Κανείς δεν αφισβήτησε φέτος τα ποσά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανείς. Και αποτείουμε εδώ φόρο τιμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντίθετα, κάποιες αντιπροσωπείες σχημάτισαν μια ανασχετική μειοψηφία και διαπίστωσαν ότι ναι, δεν αμφισβητούν τα ποσά, αλλά είτε δεν δίνονται είτε δεν επιθυμούν να καταβάλουν τα ποσά. Και το συμπλήρωμα που θα κατέβαλαν για το 2012 θα εξαρτόταν από την ευόδοση των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2013. Αυτή ήταν μια θέση που ήδη από την αρχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκρινε ως απαράδεκτη. Γιατί οι πληρωμές που έχουν γίνει και οι λογαριασμοί που έχουν δοθεί θα πρέπει να αποζημιωθούν, να πληρωθούν. Και για να επαναλάβω κάτι που είπε ο κύριος Λεβαντόφσκι, η θέση, η συμπεριφορά αυτών των κρατών μελών είναι σαν τη συμπεριφορά ενός πελάτη που πληρώνει με την πιστοτική του, αγοράζει το εμπόρευμα και σπέφτει μετά στην τραπεζά του για να διαμαρτυρηθεί για την ε, εντολή πληρωμής που έχει φτάσει στην τράπεζα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και παρά τις προσπάθειες που έγιναν και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προσπάθησε να μεσολαβήσει και παρά τις προσπάθειες της Κυπριακής Προεδρίας δεν μπορέσαμε να μεταπίσουμε αρκετές αντιπροσωπείες. ώστε να ξεκινήσουμε τη συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό του 2013. Το μόνο που καταφέραμε, και είναι σημαντικό να το σημειώσουμε και να εκφράσουμε την ευαρέσκειά μας, χάρη στην επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το μόνο που καταφέραμε είναι την ψήφα του Συμβουλίου για τον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμό 5, δηλαδή για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης ε, για τους σεισμοπαθείς της Εμίλια Ρωμάνα για 670 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε αυτό το διορθωτικό προϋπολογισμό, υπαριθμό 5, θα μπορέσουμε να το ψηφίσουμε σε λίγο. Η κατάσταση τώρα έχει ως εξής. Η διορία που προβλέπουν οι συνθήκες έχει λήξει. Οπότε μέσω στο αρχικό σχέδιο του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρείται ως απαράδεκτο, μη παραδεκτό, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να καταθέσει ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού. Αυτή την κατάσταση την αντιμετωπίσαμε για διαφορετικούς λόγους πριν από δύο χρόνια. Τότε ήταν άλλο το πρόβλημα, δεν αφορούσε τα ποσά, αλλά έχαμε, έχουμε τη βούληση και το δηλώσαμε και στο Συμβούλιο, το επιβεβαίωσαν και οι συντονιστές, το δήλωσε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι συγητές μας ήταν σαφείς. Πρόθεσή μας είναι να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση υπό τους ίδιους όρους, με το ίδιο επικοδομητικό πνεύμα και στις ίδιες προθεσμίες με αυτές που ίσχυαν πριν από δύο χρόνια. Δηλαδή, ευελπιστούμε ότι θα καταλήξουμε σε τελική συμφωνία μέχρι τα τέλη του έτους. Και μάλιστα θα ψηφίσουμε την Ολομέλεια, στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου, ώστε να ξεκινήσουμε το 2013 έχοντας ένα κοινοτικό προϋπολογισμό. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες δος, κάτι που προϋποθέτει μια αρκετά διαφορετική αυτή τη φορά μεθοδολογία από τη μέχρι τώρα και όπως και πριν από δύο χρόνια κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε το νέο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει αμέσως υπόψη τις επιθυμίες ε, και των δύο σκελών της ε, Δημοσιονομικής Αρχής. Όπως φάνηκε και από τις ψηφοφορίες, δηλαδή τις τροπολογίες και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Βέβαια, πολλές από αυτές είναι αντιφατικές. Το γνωρίζουμε, δεν είναι κάτι συνήθιστο, αλλά επειδή έχουμε συνεχείς επαφές τις τελευταίες εβδομάδες, γνωρίζουμε ότι για πολλά σημεία μπορούμε να περιορίσουμε τις διαφορές μας και να γεφυρώσουμε σχετικά εύκολα τις διαφορές μας. Το είπα πάντως και στην Κυπριακή Προεδρία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το λέω και δημοσίως εδώ. Είναι και ο Γενικός Διευθυντής παρών, οπότε μπορεί να κάνει και εκείνο τα σχόλιά του. Δήλωσε λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει ό,τι μπορεί και κυρίω οι συζητητέ, οι συνεργάτε του, ευχαριστώ θερμά και φυσικά και ο πρόεδρο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τηρήσουμε τι προθεσμίε και για να είναι βέβαιη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σχεδόν βέβαιη ότι στο σχέδιο προπολογισμού που θα καταθέσει, όπω και πριν από δύο χρόνια, θα υπάρχει ήδη μια προκαταρκτική πολιτική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών της Δημοσιονομικής Αρχής. Τώρα, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται ή έχει την ευθύνη να υποβάλει για κάποια σημεία και για κάποιες δημοσιονομικές γραμμές θέσεις που ανταποκρίνονται σε ισχυρές ε, πολιτικές απόψεις, για τις οποίες όμως γνωρίζει ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία, αλλά παρόλα αυτά κρίνει σκόπιμο να τις παρουσιάσει αυτές τις θέσεις δημοσίως, να προσυμφωνήσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδου ασυμφωνίε. Αυτό συνέβη και πριν από δύο χρόνια. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε το δεύτερο σχέδιο προπολογισμού, για το οποίο εκ των προτέρων γνωρίζαμε ότι μερικά σημεία δεν θα μπορούσαμε να τα δεχτούμε. Ήταν γνωστό και δεδομένο. Καταφέραμε όμω παρόλα αυτά να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο σε κάποιες τροπολογίες. Κάτι που μας επέτρεψε στη συνέχεια και με αυτή τη νέα βάση που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξουμε σε παρόμοια ψηφοφορία στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και να διεκπαιρώσουμε το θέμα στην πρώτη ανάγνωση, χωρίς καν διαδικασία συνδιαλλαγής. Ίσως χρειαστεί κάποιος τριμερής διάλογος για να τηρήσουμε την προθεσμία και να διακπεραιώσουμε το θέμα μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Αυτά λοιπόν. Έχουμε καταρτήσει και ένα χρονοδιάγραμμα συναντήσεων και επαφών μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Προεδρίας, τον κύριο Μαυρογιάννη, και με τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι θα έχουμε συνάντηση την επόμενη Δευτέρα. Θα έχουμε και άλλες φυσικά συναντήσεις και φυσικά και τηλεφωνικές και με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες θα έχουμε συνεχείς επαφές. Δεν ξέρω αν οι συγητές τώρα θέλουν να συμπληρώσουν την παρουσίαση αυτή. Pas Καλώς, δεν θέλω. Λοιπόν, μια που έχουμε την ε, ε, τύχη να παρευρίσκεται ο κύριος Γενικός Διευθυντής, θα μπορούσατε να μας πείτε, σας παρακαλώ, τι γίνεται από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να θυμίσω κάτι. Ο διορθωτικός προπολογισμός υπαριθμών 6 ε, για τον οποίο συζητούμε όλο αυτό τον καιρό, παραμένει επιτάπητος. Και στην παρούσα φάση θα πρέπει να αποφανθεί το Συμβούλιο Υπουργών για το σχέδιο προπολογισμού, αυτό το διορθωτικό υπαριθμό 6 και η διαδικασία που έχει αρχίσει θα πρέπει να συνεχιστεί. Θυμίζω ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό και λόγω των θέσεων που έχει λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και διότι από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υφιστάμεθα ισχυρή πίεση ε, χρονική γιατί πρέπει να καταβάλουμε αυτές τις πληρωμές. Τώρα, για το σχέδιο προϋπολογισμού, άριστα περιγράψατε ο ίδιος την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να καταρτήσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013, νέο, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί γύρω στις 23 Νοεμβρίου. Είναι πάρα πολύ σφιχτή αυτή η προθεσμία, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι όλα έτοιμα εκεί γύρω στις 23 Νοεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό. Όπως είπατε και εσείς ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος που θα έχουμε για τη διαπραγμάτευση και την επίτευξη συμφωνίας εν ώψη της έγκρισης του προϋπολογισμού στη Σύνοδο Ολομελίας του Δεκεμβρίου. Ουσιαστικά θα έχουμε την εβδομάδα που αρχίζει από την ε, Παρασκευή 23 νοεμβριου πεντε 5-6 μέρες, εκ των οποίων 5 εργάσιμες πάνω κάτω για να συμφωνήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μέθοδο εργασία. νομίζω ότι τέλεια επίσης συνοψίσατε την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούν όσο γίνεται πιο στενά τα τρία θεσμικά όργανα. Πάντα με συμβασμό στις θέσεις ο ένας άλλο, βεβαίω. Αλλά ή δυνατόν θα πρέπει κάπου να εξευρεθούν ε, σημεία ή παιδεία συνένεσης για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε το έδαφος για την επίτευξη ταχείας συμφωνίας. Αυτά ήθελα να σας πω. Συμπληρωματικά, στη δική σας παρουσίαση, Πρόεδρε, και βεβαίως μπορείτε να υπολογίζετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσήλωση και την αφοσίωσή της έτσι ώστε ο προπολογισμό του 2013 να εγκριθεί εγκαίρω και να αποφύγουμε τον εφιάλτη και τις πολύ ανητικές συνέπειες της ιστορίας των 12 τιμωρίων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια-δυο συμπληρωματικέ ερωτήσεις, αλλά ζήτησαν συνάδελφοι το λόγο. Ο κύριος Χάρτονγκ πρώτος. Πρόεδρε, μαζί με τον κύριο Σούλτς λέτε εσείς στον τύπο ότι ορισμένα κράτη-μέλη αρνούνται ε, να βάλουν το χέρι στη τσέπη για το 12. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά έχουν τους λόγους τους από τα 9 εκατομμύρια, τα 7,2 ε, είναι του Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής και των Διαρθρωτικών. Ε, Κομισιόν και Κοινοβούλιο έχουν κάνει δύο σοβαρά λάθη. Έχουν πάρει πάρα πολλές υποχρεώσεις ε, μετά από την πίεση χωρών της Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης και δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα χρήματα για τιμολόγια που εκκρεμούν, γιατί πού θα τα βρούμε τα λεφτά, πρέπει να τα πάρουμε από αλλού. Δεν φταίνε τα κράτη-μέλη που αρνούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη για επιπλέον 9 δι. Φταίνε το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν έχουν κάνει σωστά του υπολογισμού. Και ποιο την πληρώνει, ποιο είναι το κορόιδο, ο Ευρωπαίο πολίτη. Λυπάμαι πάρα πολύ για τη θέση του Κοινοβουλίου στι διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ. Καλώ κύριε Χάρτονγκ. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο διαφωνούμε λοιπόν. Εγώ είμαι υπερήφανο για τη στάση του Κοινοβουλίου. Θέλει να απαντήσει αμέσως ο Σαλβαδόρ Γκαρίγκα στα όσα άκουσε. Σε αυτή εδώ την Επιτροπή Προϋπολογισμών έχουμε μεγάλη αντοχή και αντέχουμε πολλά πράγματα να ακούμε και αυτά που δεν συμφωνούμε και που μας φαίνονται σφαλμένα. Αυτά που είπε ο κύριος Χάρτονγκ είναι πάρα πολύ βαριά, δεν είναι δικαιολογημένα και θα παρακαλούσαμε είτε να τα εξηγήσει λίγο περισσότερο είτε να τα αποσύρει αυτά που είπε. Δεν θέλει ο κύριος Χάρτον. Ο κύριος Χάρτον είναι υπερήφανο να μην πληρώνει ε, τα τιμολόγια και τους οργανισμούς που έχει υπογράψει. Θαυμάσια. Είναι ο μόνος εντός της αιθούση που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, ο Γιώραν, μισό λεπτό. Για αυτό το θέμα πάλι ακόμα όχι. Για κάτι άλλο. Λοιπόν, Άλλο θέμα. Εντάξει. Ε, ε, πρώτα όμω ο Λάσλο Σούριαν. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ να πω κάτι πιο θετικό από τη συζήτηση μέχρι τώρα. Πρώτον, πιστεύω ότι αναγνωρίζουμε ότι οι συγητές δεν ζητούν το λόγο. Σημαίνει ότι μας κάλυψε αυτό που είπατε εσείς πλήρως και τους ε, εισηγητές, άρα και εμείς θα πρέπει να τους καλύψουμε και να τους υποστηρίξουμε. Εγώ έχω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που είναι η συμπεριφορά και η τεχνική ίδια και η τακτική της Προεδρίας. Δεν συμμερίζομαι πλήρως στις δικές σας απόψεις ότι τα κράτη-μέλη είπαν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν ότι αυτά τα κράτη-μέλη που δηλώνουν αδυναμία πληρωμή ευθύνονται για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Το Κοινοβούλιο είχε μια σαφή θέση και την εξηγήσατε εσεί πολύ σαφώ την Παρασκευή και το υποστηρίξαμε εμεί στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση. Το επόμενο βήμα ποιο ήταν. Το Συμβούλιο είχε άλλη θέση. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα δεχτούν αυτά που λέμε εμεί. Και όταν έχουμε δύο σαφείς θέσει, δουλειά τη προεδρία είναι να αναζητήσει λύση για να συγκεράσει τις δύο διαφορετικές εκδοχές. Δεν υπάρχει τρίτη εκδοχή. Δεν ψηφίζουν στο Συμβούλιο. Και έχουν μια θέση που είναι τελείως αντίθετη με τη δική μας ακόμα και όταν έχεις μια τελείως αντίθετη άποψη μπορείς να βρεις ένα συμβιβασμό. Αλλά αν δεν έχεις καμία θέση από την άλλη μεριά, τι να συμβιβάσεις, το ανύπαρκτο. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα στις επόμενες διαπραγματεύσεις και στους επόμενους τριμερείς διαλόγους. Θα συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά. Δεν ψηφίζει το Συμβούλιο, δεν καταλήγει, δεν ε, αποκρισταλώνει θέση. Τι θα γίνει. Αν παραμείνει αυτή η κατάσταση, δεν πρόκειται εμεί να μπορέσουμε ποτέ να λύσουμε το πρόβλημα. Οπότε, Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να στείλουμε κάποια μηνύματα. Δεν ξέρω προς ποια κατεύθυνση και με ποιον αποδέκτη, αλλά ας πάρουν μια απόφαση επιτέλους, ας ψηφίσουν κάποια στιγμή. Και, και εμείς να δηλώσουμε σήμερα ότι είμαστε πρόθυμοι να λύσουμε το πρόβλημα και επιδεικνύουμε καλή βούληση, Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι πρέπει να πληρωθούν αυτά τα 9 δι. Μπορούμε να συζητήσουμε όμως το χρονικό ορίζοντα. Δεν είναι επιπλέον δαπάνες. Πριν από ένα χρόνο δεσμευτήκαμε, ήταν υποχρέωσή μας. Και το είχαμε ξαναπεί ότι δεν θα φτάναν τα λεφτά. Και αν μπορεί κάποιο να κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ τη ανάληψη υποχρεώσεων και των πληρωμών, δεν θα εκπλαγεί ε, να διαπιστώνει εκ των υστέρων ότι δεν φτάνουν τα χρήματα για τις πληρωμές, αλλά έχουμε αναλάβει υποχρεώσεις. Αλλά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που είναι η Δημοσιονομική Αρχή, τελικά θα πληρώσουν την ύφη. Ο τρόπος, οι τεχνικές λεπτομέρειες μπορούν να συζητηθούν. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να δείξουμε κάποια ευελιξία και όχι ακαμψία. Η ακαμψία είναι ότι θα πρέπει να πληρωθούν, γιατί το περιμένουν οι πολίτες. Τώρα τα τεχνικά, το πότε, αυτές οι λεπτομέρειες μπορούμε να τις δούμε. Κύριε Πρόεδρε, ίσως θα πρέπει να δείξετε λίγο περισσότερο ταλέντο από όσο ε, διαθέτεται ήδη που είναι τεράστιο. Ε, αλλά θα πρέπει εσείς να αναλάβετε τώρα αυτό το καθήκον για να ανταποκριθείτε σε μια ατάλλαντη προεδρία του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ για τα προσωπικά αυτά που είπατε, αλλά πολιτικά δεν συμμερίζομαι την κρίση σας βεβαίως. Η Κυπριακή Προεδρία έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες και τη χρειαζόμαστε ακόμα και την εμπιστευόμαστε. Ο Γιώραν Φέρνου. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ να συνεχίσω μετά από αυτά που είπε ο Λάσλο Σουριέν για τη φύση της σύγκρουσης που είχαμε. Εγώ έχω παρακολουθήσει 11 διαπραγματεύσεις ε, δημοσιονομικές. Αυτή είναι η 11η και ποτέ δεν είχα αυτή την εμπειρία παλιότερα. Είναι μοναδική η κατάσταση και είναι παράξενο γιατί όπως είπε ο Λάσλο το Συμβούλιο εξ αρχής ζήτησε χαμηλό επίπεδο πληρωμών ως απο, απόλυτη προϋπόθεση για μια συμφωνία για τον προπολογισμό του 2012. Αυτό είναι σαφές. Δέχτηκαν ε, βασικά το επίπεδο υποχρεώσεων κτλ. Αλλά η απόλυτη τους, ο απόλυτος όρος ήταν χαμηλό επίπεδο πληρωμών. Και τους είπαμε και εμείς εξ αρχής και τους το είπε και η Κομισιόν ότι συγγνώμη αλλά γνωρίζουμε ήδη πως αυτό τελικά δεν θα λειτουργήσει. Ωστόσο, αυτό ήθελαν οπωσδήποτε, πάση θυσία. Μπάς τελικά τους κάναμε να συμφωνήσουν για μια κοινή δήλωση που λέει ότι εντάξει, αν κάνουμε λάθος, αν έχουμε υποτιμήσει την κατάσταση, η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει διορθωτικό προπολογισμό. Αυτό εξ αρχής το συμφωνήσαμε και ξέραμε ότι θα συμβεί. Στις 10 προηγούμενες διαπραγματεύσεις οι πληρωμές είχαν θεωρηθεί ως ένα είδος τεχνικό αυτόματο αποτέλεσμα των υποχρεώσεων. Εφόσον αναλαμβάνεις μια υποχρέωση, η φύση αυτή είναι ότι φτιάχνεις, συνάπτεις μια σύμβαση. Κάνεις κάτι που σε υποχρεώνει νομικά να πληρώσει του λογαριασμού σου. Άμα φτιάξει ένα σπίτι, ας πούμε, αρχίζει το χτίζει. έχεις κόσμο, χτίστες, οικοδόμου ε, εργολάβου και μετά στο τέλο λες, α, συγγνώμη, λάθος, δεν έχω αρκετά. Μα δεν πάει έτσι. Αυτή είναι η θέση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αν τα κρατημέλη θέλουν να μειώσουν τον προπολογισμό, αν θεωρούν ότι ο προπολογισμό τη Ένωση είναι πολύ μεγάλο, θα πρέπει να το κάνουν μέσα από διαπραγματεύσει και θα πρέπει να το κάνουν από πλευρά υποχρεώσεων. Γιατί αυτέ είναι το σημάδι για να προχωρήσουμε με projects και με, ε, ε, και με διαγωνισμού κτλ. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνω, αλλά αν θέλουν να το κάνουν πρέπει να ασχοληθούν με τις υποχρεώσεις και όχι με τις πληρωμές. Και ερώτηση προς την ε, Κομισιόν τώρα. Καταρχήν, αν συμμερίζω την άποψή μου. Και δεύτερον, εγώ ανησυχώ τώρα ότι ακόμα και αν λυθεί η κατάσταση όσον αφορά στο σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 6, θα καταλήξουμε σε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα το 2013. Διότι μπορούμε να δούμε ότι μια από τις θέσεις του Συμβουλίου είναι να μειώσει τις πληρωμές και για το 2013. Και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Είδαμε συμβιβαστική πρόταση, δεν ξέρω αν έχει δημοσιευθεί, εγώ ατύπως πάντως την είδα, δεν θα αναφέρω νούμερα, αλλά είδαμε μια συμβιβαστική πρόταση από την Κομισιόν που νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χαμηλή όσον αφορά τις πληρωμές για το 2013. Τι κάνουμε λοιπόν για να αποφύγουμε να καταλήξουμε στην ίδια κατάσταση το 2013 και η Κομισιόν μπορεί να πει δύο λόγια για τις ανάγκες πέρα από το σχέδιο διευθυντικού προϋπολογισμού 6 για το 12 και για το 13. Ευχαριστώ. Έιντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να είμαι ειλικρινής, έχω σιγά σιγά την αίσθηση ότι είμαστε σε ένα έργο επιστημονικής φαντασίας. Γιατί θα πρέπει λέει, να δικαιολογήσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου εξηγώντα τα κράτη μέλη ότι πρέπει να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Όταν ήρθα στο Κοινοβούλιο ποτέ δεν το είχα φανταστεί ότι θα έπρεπε να κάνω κάτι τέτοιο. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν κάποιε υποχρεώσεις και κάνουν κάποια έργα, κάποια προγράμματα, χρηματοδοτούν ή ε, προκυρήσουν διαγωνισμούς και μετά θα πρέπει να πληρώσουν και πρέπει δηλαδή να έρθει το κοινοβούλιο να εξηγήσει γιατί να το κάνουν. Απίστευτα πράγματα είναι αυτά. Εν πάση περιπτώσει, για το τι μέλη γενέστε και πολύ προσεχώς μάλιστα εντός του μηνός που θα πρέπει να ε, δουλεύουμε πραγματικά υπό μεγάλη πίεση. Πριν από δύο χρόνια όταν έγινε αυτή η συμφωνία, σε χρόνο ρεκόρ καταφέραμε να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει ένα προπολογισμό. Ε, που ήδη είχε συμφωνηθεί και ήταν πολύ γρήγορε οι διαδικασίε. Αλλά φέτο δεν είναι ακριβώ η ίδια κατάσταση, διότι φέτο δεν καταφέραμε να καθίσουμε να συζητήσουμε για τον προπολογισμό του 2013. Διότι βάζαμε ω προοπαιτούμενο ότι το Συμβούλιο θα συμφωνούσε για το διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 6. Είναι αρκετά λογικό δηλαδή να μην αρχίσουμε να συζητάμε για το επόμενο έτος χωρίς να έχουμε λύσει του φετινού τον προπολογισμό. Γι' αυτό δεν προχωρήσαμε στις πραγματεύσεις. Ελπίζω αυτό να γίνει και σίγουρα από πλευρά κοινοβουλίου θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε σε συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να επαναλάβω τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς δεν αλλάξαμε θέση σε ό,τι αφορά την πρόταση τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε αλλάξαμε θέση ειδικά στις πληρωμές Τίποτα καινούριο δεν υπάρχει, ούτε νέες ε, προοπτικές, προβλέψεις, στοιχεία, καμία διαπραγμάτευση. Και οι πληρωμές που υπερασπίζεται το Κοινοβούλιο και θα πρέπει να είναι στην πρόταση της Επιτροπής, θα πρέπει να είναι το ίδιο ποσό που προτινόταν για το 2013. Γιατί το λέω αυτό. Διότι στο τελευταίο έγγραφο που μας παραδόθηκε την περασμένη Παρασκευή, στο τέλος της συνδιαλλαγής, εμφανίστηκε μια αλλαγή, η πρόταση αλλαγή για το επίπεδο πληρωμών. Και το επίπεδο ήταν αυτό που πρότεινε το Συμβούλιο συν 1,4 δις. Αυτό δεν είναι αύξηση στις πληρωμές, αλλά είναι μεταφορά ενός τμήματος του υπαριθμών 6 ε, των λεγόμενων ε, suspended claims στο επόμενο οικονομικό έτος. Μην κάνουμε λάθος εκεί και γίνουν τίποτα αλχημίες με τα ποσά και να χάσουμε τη θέση μας και τον ορίζοντά μας. Η πρώτη πρόταση που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληρωμές είναι αυτή που χρειάζεται να ε, καταβληθεί. Και θυμίζω ότι όταν έκανε την πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας θύμισε ότι η πρόταση βασιζόταν στο γεγονός ότι το 2012 είχε κλείσει και ε, είχε καλυφθεί πλήρω και από πληρωμέ. Δεν ξανανοίγει αυτό. Γιατί με το διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 6 πληρώνουμε τα τιμολόγια μόνο μέχρι 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή, Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα εκκρεμούν και θα πρέπει κάποτε να καταβληθούν εντός του 13. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να προσθέσω, και ήδη ακούστηκε, είναι αυτές οι περίφημες δηλώσεις οι γραπτές για τις συμφωνίες που κάνουμε λέει με το Συμβούλιο. Γιατί και αυτό είναι λίγο επιστημονική φαντασία. Τελικά υπογράφουμε ένα χαρτί με το Συμβούλιο που δεσμευόμαστε να τηρούμε το νόμο. Και όχι μόνο το νόμο, αλλά και τα συμφωνηθέντα που λέει το έγγραφο. Οπότε πώς μπορούμε εμείς μετά να διαπραγματευτούμε τον προπολογισμό για το 2013 δεν θα πρέπει να ξαναπέσουμε στην ίδια παγίδα και να κάνουμε το ίδιο σφάλμα, δηλαδή να υπογράψουμε ένα έγγραφο που δεσμεύεται το Συμβούλιο να μελετήσει, λέει, αλλαγέ στον προπολογισμό σε περίπτωση που χρειαστεί. Όπω λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξαντλείται ο προπολογισμό, δεν έχουμε λεφτά για να βγάλουμε το έτο και το ε, Συμβούλιο εξακολουθεί να αρνείται ε, την έγκριση του διορθωτικού προπολογισμού θα βρούμε μπροστά μας τα προβλήματα. Δεν μπορεί το Συμβούλιο να εγκρίνει αυτά τα κονδύλια για να τελειώσουμε τη χρονιά. Και γιατί να πιστέψουμε ότι το 13 θα αλλάξει θέση του. Εγώ δεν εμπιστεύομαι καθόλου πια το Συμβούλιο. Ευχαριστώ και τελείωσα αυτά. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Σημαντική συζήτηση. Έχω μακροσκελή κατάλογο μιλητών. Σας παρακαλώ να είστε ακριβείς και συνοπτική στα σχόλιά σα. Δεν πρόκειται να επαναλαμβάνουμε τώρα όλη τη γνωστή επιχειρηματολογία. Τα ακούσαμε και στη συνδιαλλαγή. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Α περιοριστούμε λοιπόν στο απολύτω απαραίτητο. Κυρία Αντρέασεν. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με ότι θα πρέπει να πληρωθούν οι λογαριασμοί, αλλά Ακόμη σε οποιοδήποτε οργανισμό του κόσμου, για να πληρώσει κανείς τα τιμολόγια, πρώτα ελέγχει αν ε, έχουν ε, ε, παραδοθεί τα αγοραστέντα ή έχουν τελεστεί οι υπηρεσίες. Και αυτό με ανησυχεί, γιατί δόθηκαν τιμολόγια και απαιτούνται δαπάνες από τα Υπουργεία για να κρατηθούν τα κονδύλια που προέβλεπε το πολιτής δημοσιονομικό πλαίσιο. Ναι, πρέπει να πληρώσουμε τα τιμολόγια, να πληρώσουμε του λογαριασμού, αλλά είναι πραγματικοί αυτοί οι λογαριασμοί. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι αυτά τα τιμολόγια που ζητούν τα κράτη-μέλη, οι διάφορε διοικήσει είναι πραγματικά. Και νομίζω ότι θα ξεσηκωθούν οι διάφοροι τομεί, είπαμε, να ζητούν τα κονδύλια. Αλλά δεν βλέπω κανένα να έχει ξεσηκωθεί σε κανένα κράτο μέλο για τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που βλέπω είναι να ξεσηκώνονται πολύ στα κράτη-μέλη κατά των μέτρων λιτότητας. Βλέπω στην Ισπανία να πηδούν άνθρωποι από τα παράθυρα ε, διαμαρτυρούμενοι για τις εξώσεις. Πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα Αέρασμος, κύριε Λαμασούρ και αγαπητοί συνάδελφοι. Όχι, αδιαφορούν πλήρως. Ανησυχούν πολύ περισσότερο για άλλα πράγματα. Έχουν άλλες έγνοιες. Εμάς μας προβληματίζουν αυτά τα χρήματα, αλλά τα χρήματα αυτά μπορεί να τα χρειάζονται τα κράτη-μέλη για εσωτερικού σκοπού και θα πρέπει να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν όντω αυτά τα κονδύλια για εσωτερικού σκοπού. Κυρία Ανδρέασε, έχουμε αυτή την αίθουσα πολύ πιο αρμόδιους από εσά και από μένα για να μιλήσουν για την Ισπανία. Μερικές χώρες, όπως και η δικιά σας, αρνούνται να καταβάλουν 1,47 δις, περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δηλαδή, που οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ισπανία μόνο για λογαριασμούς και τιμολόγια για τα οποία δεν αφισβητείται από την Ηνωμένα Βασίλειο τίποτα. 1,8 δις ε, για την Ιταλία θα πρέπει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει στην Ιταλία. 1,5 ε, δις θα πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψει, να αποζημιώσει την Πολωνία για ανηλυμένους ε, υποχρεώσεις και για καταβληθέντες λογαριασμούς. Γιατί μερικοί θα πούνε ότι είναι οι χώρε του Club Med, δεν είναι σοβαρέ χώρε. Να πάρουμε μια σοβαρή χώρα. Η Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει στη Γερμανία 869 ε, εκατομμύρια. Αυτή είναι η κατάσταση. Και Δύο φορές ρώτησα τους υπουργούς. Ήταν παρόντες οι υπουργοί, όχι ε, υπάλληλοι. Ήταν εκεί οι υπουργοί και τους ρώτησα για τα 9 δισεκατομμύρια. Αμφισβητεί κανείς τα τιμολόγια, αμφισβητεί κανείς τους λογαριασμούς, κανείς. Κανεί υπουργό δεν αμφισβήτησε τίποτα. Πέρυσι υπήρχαν αμφισβητήσει. Φέτο κανένα δεν αμφισβήτησε αυτά τα ποσά. Κύριε Ανδρέασεν, η φετινή κατάσταση δείχνει ότι παρά την πρόοδο που σημειώσαμε σε ό,τι αφορά την εξακρίβωση της γνησιότητας των τιμολογίων και το γεγονός ότι είναι αδιάψευστα τα ποσά που περιλαμβάνουν, είναι ότι παρόλα αυτά έχουμε μία κρεμή διαδικασία. Και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί και στην τελική συμφωνία μας και θα το συζητήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνεδρίαση των συντονιστών και στην ε, Επιτροπή μας, στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών, η, Συντο... η Συντόνια. Όντως, η εμπειρία τη διαλλαγής ε, και της παρασκευή και τη Τρίτη ήταν απογοητευτικέ, γιατί δεν κατέστη δυνατό να ακούσουμε καμία πρόταση από το Συμβούλιο. Ήμασταν εκεί, αλλά συζήτηση δεν μπορούσε να γίνει, γιατί το Συμβούλιο ήταν ανίκανο να υποβάλει οποιαδήποτε πρόταση, να παρουσιάσει οποιαδήποτε θέση. Οπότε με εικασίες χρειάστηκε να δουλέψουμε. Δεν μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε και θα ήθελα πραγματικά να εξάρω τις προσπάθειες του Προέδρου και των δύο εισηγητών που πήγαν στο Συμβούλιο είτε το απόγευμα της Τρίτης και σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από το Συμβούλιο. Πήγατε για να διευκρινίσετε τη θέση, αλλά δεν υπήρξε καμία θέση του Συμβουλίου, καμία θέση ειδική πλειοψηφία. Έστω και παράδεκτη. Δεν είχαμε τίποτα να στηριχθούμε. Δεν ήταν διάλογο ουσιαστικά. Απλώ καθόμασταν και προσπαθούσαμε να μαντέψουμε τι ζητά το Συμβούλιο. Κατά τη γνώμη μου, ήταν πολύ δυσάρεστη και καθόλου ικανοποιητική η μέθοδος εργασίας. Τώρα έχουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, κατάσταση τη σημερινή. Γιατί λέμε να λύσουμε το πρόβλημα για τις ακρεμείς πληρωμές για το 2012 και τον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 6. Και φυσικά για τους λόγους που ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Ένα επιπλέον θέμα όμως θα πρέπει να εξεταστεί επίσης. Η σημερινή κατάσταση προκλήθηκε από κάτι που πολλοί πέστε του όπως θέλετε, ευρωσκεπτικιστέ, απλώ σκεπτικιστές, δεν μπορούσαν να φανταστούν. Ότι δηλαδή η εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων θα ήταν τόσο πετυχημένη, τόσο καλή. Γιατί ο προπολογισμό γίνεται χρόνια ολόκληρα. Έχουμε πολύ χαμηλότερα, είχαμε στο παρελθόν πολύ χαμηλότερα επίπεδα πληρωμών από τα επίπεδα ανάληψη υποχρεώσεων. Γιατί θεωρούσαμε ότι σε μεγάλο βαθμό τα προγράμματα θα αποτύχουν και ότι δεν θα μπορέσουν οι δικαιούχοι να αξιοποιήσουν τα κονδύλια. Τα τελευταία όμως τρία-τέσσερα χρόνια είχαμε μια κατάσταση για την οποία δεν ήμασταν προετοιμασμένοι και από ό,τι φαίνεται ακόμη τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να χωνέψουν αυτή την αλλαγή. Ότι δηλαδή όντως είναι επιτυχημένα τα προγράμματα και ότι έχουν εκπαιδευτεί, έχουν μάθει από την εμπειρία οι δικαιούχοι και μπορούν να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν αυτά τα κονδύλια. Και μας, μας λείπουν πιστώσεις πληρωμών που να ανταποκρίνονται στη νέα πραγματικότητα. Αυτή είναι η νέα κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την οτροπία μας για να αντιμετωπίσουμε τη νέα πραγματικότητα με που δείχνει μια επιτυχία των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν την εκκρεμότητα από το 2012, αλλά να μην ξεχνάμε ταυτόχρονα ότι έχουμε μπροστά μας και τον προϋπολογισμό του 2013. Και εδώ έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν μας υποβληθεί το νέο σχέδιο προϋπολογισμού, θα πρέπει να φροντίσουμε το σχέδιο προπολογισμού του 2013 να είναι όσο πιο ρεαλιστικό γίνεται για να αποφύγουμε παρόμοια κατάσταση του χρόνου τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Εγώ δεν πιστεύω ότι η πίεσή μας για το 2012 θα πρέπει να μας απαλλάξει από εξίσου σκληρή εργασία για το 2013. Και έχω και άλλη ε, συγκεκριμένη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την γενική μεταφορά μετά τις καθερινές διακοπές. Δεν θυμάμαι, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πότε ήταν. Ρώτησα τότε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι περισσότερες από τις πληρωμές που ακυρώθηκαν, που ήταν η πηγή των πιστώσεων πληρωμών, δεν ήταν για προγράμματα που είχαν αποτύχει ακυρωθεί, αλλά οφειλόταν σε αναβολές. Έχουν συμπεριληφθεί αυτά στον προϋπολογισμό, έχουν ενταχθεί πια ή θα αναβάλλονται παόριστον. Ή χρειαζόταν ένας χρόνος αναμονής για τις λεπτομέρειες των συμβάσεων, αλλά κάποια στιγμή, την άνοιξη το καλοκαίρι, θα υποβληθούν αυτές οι ε, απόλυτα εύλογες ε, απαιτήσει. Τα λαμβάνετε αυτά υπόψη, έχουν μπει στον προπολογισμό αυτές οι αναβολές. Και επίση, ε, τι γίνεται με την συμβαστική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που είδαμε την Παρασκευή. Εξαφανίστηκε. Και τώρα, η πρόταση να εξετάσουμε ένα διορθωτικό προπολογισμό για το 2013 σε νωρίτερο στάδιο θα εμφανιστεί κάποια στιγμή. Αλλά δεν ξέρω αν αυτή η λύση είναι ρεαλιστική και εφικτή. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος δεν ε, ήθιστε ε, να εξετάζουμε διορθωτικούς προϋπολογισμούς ε, νωρίς μας τον χρόνο. Θα ασκηθεί πίεση βέβαια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανακατανομή. Βέβαια, αν υπάρχει δυνατότητα ανακατανομή, θα πρέπει να γίνει. Αλλά, και τελευταία ερώτηση προς την Επιτροπή. Ποια θα είναι τα ασθενή τμήματα της πολιτικής που θα είναι τα θύματα αυτής της ανακατανομής. Από πού θα πάρετε τα κονδύλια στις αρχές του 2013 ή μόπως θα είναι μια ε, ιονή χειρονομία. Γιατί ενα τέτοιο, ένα τέτοιο σχέδιο προπολογισμού σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υλοποιηθεί στις αρχές του 2013. Ευχαριστώ Σιδωνία, εξαιρετική συζήτηση. Πολύ συγκεκριμένη και πολύ κέρια. Ο κύριος Γκοντμάνης. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο. Καταρχήν πιστεύω πως είμαστε σε μια κατάσταση όπου ο προπολογισμό που εγκρίναμε το 2005 το Δεκέμβριο, όταν δηλαδή δεν υπήρχε κρίση στον ορίζοντα, το πρόβλημα είναι ότι ο αντίκτυπος της κρίσης έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Κανονικά, σε εθνικό επίπεδο, οι προπολογισμοί διορθώνονται, όμως η κατάσταση επιδεινώνεται. Και αυτό τώρα δοκιμάζεται γιατί έχουμε μια πλειοψηφία, μια πλειοψηφία που κάθε χρόνο μπλοκάρουν, περιορίζονται οι πληρωμές, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε προϋπολογισμό διαφορετικό από ό,τι τα κράτη. Αν είχαμε τον προϋπολογισμό για του χρόνου, θα έπρεπε να έχουμε και κάποιο μηχανισμό για να βγούμε, γιατί φαίνεται σαν να μπορούμε να αλλάξουμε κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό, αλλά δεν γίνεται αυτό και στο τέλος έχει πρόβλημα. Δεύτερον, το πρόβλημα από ό,τι κατάλαβα εγώ είναι ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε συμβιβασμό. Όλοι έχουμε άποψη. Στη συνοχή έχουμε 9 εκατοδείς, τα χρήματα που έχουμε όμως ε, είναι 3 ε, εκατομμύρια. Άρα μας λείπουν 6 δις. Για τα προγράμματα ανάπτυξης υπαίθρου, από τα 3 δις, μόνο 2 δις είναι διαθέσιμα. 35% δηλαδή λείπει από την Κομισιόν. Αν είναι περίπου αλήθεια ότι κάποια φάση ήταν έτοιμη μια συμφωνία για 1,4 δις που θα αφαιρεθεί από το διευθυντικό προϋπολογισμό, πράγμα που ήταν ίσως θέση του Συμβουλίου, θα παρότρινα την Επιτροπή να, το, να, να, να τα βολέψει έτσι. Γιατί αν δεν εγκριθεί τίποτα, τελικά θα έχουμε προβλήμα, πρόβλημα και θα τα σπρώξουμε όλα στο MFF και θα πληρωθούν μόνο τα χρέη. Το καλό είναι ότι στη συνοχή και στην ανάπτυξη πέθρου οι δικαιούχοι δεν έχουν υποφέρει, διότι όλα αυτά πάνε στον προπολογισμό της κυβέρνησης και στο έλλειμμά τη γιατί οι δικαιούχοι πρέπει να πληρωθούν ούτως ή άλλως. Είτε δώσει αποζημιώσει η Ευρώπη είτε όχι. Το πρόβλημα είναι όμως ε, είναι ότι δημιουργείται φαύλο κύκλος, γιατί αν δεν πληρωθούν από την Ευρώπη ε, δημιουργούνται ελλείμματα στους εθνικούς προπολογισμού. Τι έχω να προτείνω εγώ όμως στην Επιτροπή. Αλλά κοιτάξτε προσεκτικά, κοιτάξτε προσεκτικά τον διορθωτικό προπολογισμό. γιατί για τη συνοχή έχουμε γνώση και, ανταγωνιστικ... και σύγκληση. Σύγκληση και ανταγωνιστικότητα. Στη σύγκληση όμως είναι οι φτωχότερες χώρες και αυτή οι, αυτές οι περιοχές ε, παραμένουν οι περιοχές μεταβατικές περικόπτονται κατά 25%, οι ανταγωνιστικές κατά 10%, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Παρακαλώ, Πρόεδρε, πρέπει να βρεθεί η τροπολογία ε, συμβιβαστική, γιατί δεν καταλαβαίνω. Αν είναι θέμα 1,4 δις, εμείς πολύ ευχαριστώ θα θέλαμε χρήματα στη χώρα μου, αλλά, αλλά το βασικό είναι να βρούμε συμβιβαστική. Γιατί αν δεν βρεθούν έστω αυτά τα χρήματα, στο τέλος δεν θα πάρουμε τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομο θα είμαι, γιατί ξέρω ότι ανησυχείτε για το χρόνο και έχουμε και πολλά θέματα να διεκπαιρεώσουμε. Αλλά αισθάνομαι την υποχρέωση καταρχά να αντιδράσω σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Ανδρέασεν. Γιατί ειλικρινά μένω εμβρόντιτος. Δεν καταλαβαίνω σε τι αποσκοπεί η κυρία Ανδρέασεν με αυτά που λέγει. Διότι τι μιλάει για πλαστά τιμολόγια, δηλαδή για μια διοίκηση που δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο, ειλικρινά σας το λέω. Δηλαδή, τι επιχείρημα είναι αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς ε, τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, να πει ότι οι υποχρεώσεις που έχουμε ε, δεν είναι σωστές, δεν ευσταθούν. Θα παρακαλούσα την κυρία Ανδρέασεν ε, για λόγους σεβασμού της ε, αλήθειας και με σεβασμό ε, απέναντι σε ανθρώπους που ζουν τραγωδίες να μην ρίχνει τέτοιες σκιές υποψίας για τα τιμολόγια και τη διοίκηση. Επίσης, για τα όσα είπε ο Λάσλο για το ρόλο της Προεδρίας. Εσείς, Πρόεδρε, ξέρω ότι έχετε ένα θεσμικό ρόλο και μια υποχρέωση να προσπαθείτε να ενθαρρύνετε την Προεδρία να βρει κάποια λύση. Προεδρία του Συμβουλίου. Αλλά εφόσον υπάρχει αντίφαση στο εσωτερικό του Συμβουλίου το ίδιο, όταν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, γι' αυτό το λόγο υπάρχει Προεδρία, για να προσπαθεί να βρει μια πρόταση που να ακυρώνει τις ίδιες τις αντιφάσεις στις εσωτερικές του Συμβουλίου. Εξ όσων γνωρίζω, μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει αυτό η Προεδρία. Έχουμε ένα πρόβλημα πληρωμών, όχι ανάληψη υποχρεώσεων, που είναι εικονικό το πρόβλημα και είναι πιο εύκολο να συμφωνήσει. Για πληρωμέ πρόκειται τώρα. Παρακαλώ Πρόεδρε, σας ενθαρρύνω με τη σειρά σας εσείς να παροτρύνετε την Προεδρία να προσπαθήσει να αποκρισταλώσει μπας περιπτώσει μια κοινή θέση στο Συμβούλιο για να δούμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ φίλε μου, λέει ο Πρόεδρος, ο Γιάννη Μόλντορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σύντομα και γρήγορα το κλειδί για τη λύση παραμένει ε, το σχέδιο του διορθωτικού προπολογισμού. Πέρσι συμφωνήσαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νέα ποσά χρειαστεί και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να τα μελετήσουν σοβαρά για να συμφωνήσουν. Αυτό δεν έγινε το Συμβούλιο θα πρέπει να τιμήσει τις υποσχέσεις τους και να το, το υπενθυμίσουμε. Όταν έρθει η λύση για τον ε, ε, διορθωτικό προπολογισμό των παριθμών 6 και τιμήσει τις υποσχέσεις στο Συμβούλιο, τότε θα αρχίσουμε να συζητάμε για το 13 και να είναι με ε, αρκετή ανάληψη υποχρεώσεων για να μπορέσει να καλύψει τις πληρωμές και ίσως χρειαστεί και το 13 μια νέα λύση τέτοια. Αλλά η λύση θα έρθει από τον τάμπ υπαριθμών 6. Μάλιστα. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να προσθέσω εγώ μερικά σχόλια. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα τώρα οργανωτικής φύσεως. Με τους, σύντονις με τους ε, εισηγητές, συγγνώμη. Τζοβάνι και Φραντσέσκα. Έχετε προβλέψει από ό,τι ξέρω ε, συνεδρίαση εργασίας με την Κομισιόν και την Προεδρία τώρα. Αλλά πρέπει και να ψηφίσετε. Λοιπόν, τι να κάνουμε, να περάσουμε στι ψηφοφορίε, θα σα προτείνω, θα πω δύο λόγια πρώτα. Ε, θα ψηφίσουμε τον πέμπτο διορθωτικό προπολογισμό δεδομένη τη σημασία που έχει για σας, ε, ε, του Ιταλούς εισηγητέ. Και μετά διαλέξτε, θα μείνετε για τις υπόλοιπες ψηφοφορίες ή θα πάτε στη συνεδρίασή σας. Δουλεύουμε όπως η Βουλή των Κοινοτήτων. Αν χάσουμε ένα αριστερό και ένα δεξιό βουλευτή ταυτόχρονα, πολιτικά έχουμε ισορροπία και μπορείτε να μην ψηφίσετε κιόλα. Δεν τρέχει τίποτα. Συμφωνείτε? Ωραία. Λοιπόν, τελειώνω απλώς τη φράση μου. Ευχαριστώ όσους ε, μίλησαν για αυτό το θέμα και θέλω να πω το εξής. Απευθύνω στον κύριο Γενικό Διευθυντή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως μας επιβεβαιώσατε, από τώρα ήδη εργάζεται για το νέο σχέδιο προϋπολογισμού. Έχουμε όλοι συμφέρον να ε, καταλήξουμε στο προπέρσινο αποτέλεσμα. Δηλαδή ένα σχέδιο προϋπολογισμού που θα το έχουμε τόσο πολύ δουλέψει και προετοιμάσει όλοι μαζί, ε, ώστε γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι θα το εγκρίνουν οι πάντες όπως είπατε πολύ σωστά, ο καθένας ε, διατηρώντας τις θεσμικές του ευθύνες. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει ή άλλες που θεωρεί ότι οφείλει να τις υποβάλει γνωρίζοντας ε, ότι δεν θα δοθεί συνέχεια. Μπορεί να προκύψει αυτό βάσει των ευθυνών της Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων για να ξέρουμε ποια θα είναι τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν ε, για να μην ε, επιβραδυνθεί συνέχεια των εξελίξεων από πλευρά Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Τώρα πρέπει να σας πω ότι για το Κοινοβούλιο, το είχα πει και στον τριμερή διάλογο της Δευτέρας και το επαναλαμβάνω δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Προπολογισμών. Το έγγραφο που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το non-paper, εν πάση περιπτώσει, το συμβιβαστικό, την περασμένη Παρασκευή, ε, το βράδυ, είναι ένα έγγραφο που μας αποτελεί βάση εργασίας. Αυτό το non-paper το δεχόμαστε ως βάση εργασίας. Δεν δεχόμαστε τα πάντα βέβαια, δεν τα εγκρίνουμε στο σύνολό του, αλλά το θεωρούμε βάση εργασίας. Δεν ξέρω το Συμβούλιο τι φρονεί, αλλά το Κοινοβούλιο το θεωρεί βάση εργασίας. Λοιπόν, αν ξαναρχίσετε από την αρχή την κατάρτιση του προϋπολογισμού, βασιζόμενοι σε αυτό το έγγραφο ως αφετηρία και αναφορά για μας είναι απολύτως αποδεκτό. Αλλά αυτό τι σημαίνει αν εκινήσουμε από το έγγραφο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βασιστεί σε αυτό το έγγραφο, όχι στο αρχικό της σχέδιο. Γιατί κάπου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι από το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τη σήμερα ημέρα έχει μεσολαβήσει μια σειρά εξελίξεων. Όλες οι τροπολογίες του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και οι συζητήσεις που έχουμε με τα αποτελέσματά τους. Επιμένω επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγοντας ότι δεν θα πρέπει στο εσωτερικό της Κομισιόν να υπάρχει παραμικρή αμφιβολία για την αξιολόγηση αυτών που κοινώς ονομάζουμε τιμολόγια. Αν πρέπει να γίνουν αλλαγές σε σχέση με τον συμπληρωματικό και διορθωτικό προϋπολογισμό, υπαριθμών 6, αυτό θα πρέπει να είναι διόρθωση προς τα πάνω μάλλον γιατί τα 9 δις ήταν ένα υπολογισμό πριν από λίγε εβδομάδες και στο μεταξύ έχουν φτάσει και άλλα τιμολόγια. Οπότε έρχομαι τώρα να πω το εξή προς το Συμβούλιο και ευχαριστώ την Προεδρία που παρευρίσκεται. Όπως είπε ο κύριος Ζαν Ζαν, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 6 πρέπει πρώτα να εξεταστεί από το Συμβούλιο, το οποίο θα το εγκρίνει, θα το απορρίψει, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χαθεί χρόνος διαδικαστικά εκεί, για να μην υπάρξουν ολιγορίες και καθυστερήσει, ακόμα και όταν επιτευχθεί πολιτική συμφωνία, δηλαδή να μην κινδυνεύει ε, η ψήφιση του πακέτου και του προπολογισμού 2013 χρονικά. Και θα ήθελα να πω και πάλι ενώπιον της Επιτροπής Προπολογισμών παρουσία του Συμβουλίου, κάτι που γνωρίζει η Κυπριακή Προεδρία και δυστυχώς το υφίσταται όπως και εμείς. Τώρα έχουμε πρόβλημα για αυτό το θέμα που δεν είναι πολιτικό πρόβλημα που φέρνει αντιμέτωπο το Συμβούλιο για τα κράτη-μέλη. Ούτε πλέον είναι τεχνικό το πρόβλημα αξιολόγησης του ποσού και υπολογισμού του ποσού των τιμολογίων που πέρσι ακόμα έφερνε αντιμέτωπο Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόβλημά μας τώρα είναι καταρχήν, μάλλον ξεκίνησε ως τεχνικό, αλλά που μπορεί να εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό πρόβλημα μεταξύ των κρατών μελών. Έχουμε πλέον πρόβλημα των κρατών μεταξύ τους. Ορισμένα δεν αμφισβητούν την πραγματικότητα των αριθμών, ε, αυτή τη στιγμή έχει ελέγξει τα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θεωρούν ότι μερικέ χώρες το παρακάνουν στην αποστολή τιμολογίων. Ε, και αυτή η κατάσταση δεν είναι αποδεκτή, δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Εμείς τι προσπαθούμε να καταδείξουμε. Αυτό που σημαίνει, όχι για να φέρουμε αντιμέτωπα μεταξύ τους τα κράτη-μέλη, αλλά για να απευθύνουμε μια προειδοποίηση. Αν εξακολουθήσει αυτή η εμπλοκή, εάν, επαναλαμβάνω, εξακολουθήσει αυτή η εμπλοκή, εγώ θα κάνω αυτό που δεν θέλησα να κάνω μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα πω. Λοιπόν, Υπάρχει ΑΒ χώρα που αρνείται να πληρώσει την ΑΒ δαπάνη, το τάδε ποσό, ε, στη δίνα άλλη χώρα. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Δύο λοιπόν πρακτικά συμπεράσματα οφείλουμε να εξαγαγούμε από αυτή την πραγματικότητα. Κανεί δεν θέλει να συνεχίσετε αυτή η κατάσταση, ούτε η πρώτη κατηγορία κρατών, ούτε η δεύτερη. Λοιπόν, δύο είναι τα συμπεράσματα που βγάζουμε αυτή τη στιγμή βρούμε την πολιτική συμφωνία και άμεσα θα πρέπει να βελτιώσουμε τη διαδικασία μας, να ελάβουμε πιστοποίηση των ε, τιμολογίων που να είναι απολύτως πλέον αναμφισβήτητη σε κάθε χώρα συμπεριλαμβανομένων των χωρών που εμφανίζουν τον εαυτό τους ως πιο σοβαρές από τις άλλες. Και δεν μπορούν ε, τα ίδια τους τα τιμολόγια να ε, εξακριβώσουν και να επαληθεύσουν. Και μιλώ για τη χώρα μου. Γνωρίζω και άλλες, αλλά δεν έχω το δικαίωμα να τις αναφέρω και δεν είναι όλες νότιο-ευρωπαϊκές. Και το δεύτερο συμπέρασμα έχει σχέση και με το PDP ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό θα πρέπει να χρηματοδοτείται από ιδίου πόρους. Γιατί όσο είμαστε στο έλεος της κρατικής χρηματοδότησης θα έχουμε το πρόβλημα οξύτερο. Όσο η κρίση ε, βαθαίνει τόσο θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα και θα έχουμε μια κρίση μεταξύ των ε, φορολογουμένων των χωρών που είναι καθαροί συνεισφορείς με τους πολίτες της χώρες που είναι καθαροί αποδέκτες. Και θα έχουμε τα κράτη-μέλη σφοδρά αντιμέτωπα το ένα ε, απέναντι στο άλλο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Κύριε Γενικέ, Διευθυντά, θέλετε να δώσετε κάποιες απαντήσεις σε ερωτήσεις που έγιναν από μερικά μέλη της Επιτροπής Συντονία και ενδεχομένως να σχολιάσετε και άλλα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Ε, Τέθη μια ερώτηση του κυρίου Φέρμου για την κατάσταση 2013 σε σύγκριση με το 2012. Εγώ δεν μπορώ παρά να επαναλάβω τα όσα βάλαμε στην εισαγωγή του σχεδίου προπολογισμού. Ζητούσαμε το αίτημά μας πιστώσεων πληρωμών για 138 δις ξεκινούσε από την προπόθεση του σύνολου των πληρωμών του 12 θα είχαν εξασφαλιστεί. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Γνωρίζετε την κατάσταση τόσο καλά όσο και εγώ και μπορείτε να συμπεράνετε τα υπόλοιπα. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση της Σιδόνια για τις ε, γενικές ε, μεταφορές, ε, τα συνολικά εμβάσματα. Όχι, δεν θέλουμε απλά να αναβάλουμε. Φυσικά οι γραμμές για τις οποίες είχαμε προβλέψει ε, συγκεκριμένα κονδύλια και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλήρω, είναι γραμμές για τις οποίες θα πρέπει να τα πληρώσουμε κάποια, ε, κάποια στιγμή αργότερα. Αλλά και για τις γραμμές που έχουμε κονδύλια που έχουν χρησιμοποιηθεί έχουμε ε, πληρωμές που είναι ψηλότερε από αυτές που περιμέναμε και αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται σε κάθε προπολογισμό. Είναι κάτι, είναι ένας μηχανισμός που κατά κάποιο τρόπο αυτοεξισορροπείται, θα έλεγα. Δηλαδή υπάρχουμε, το, κάνουμε τον προπολογισμό για συγκεκριμένες δαπάνες και αντισταθμίζουμε με την πρόβλεψη κάποιων άλλων. Ε, ε ξεκινάμε με αυτή την ε, προϋπόθεση ότι υπάρχει μια κάποια ισορροπία και θα ήθελα να πω ότι το γενικό έμβασμα αυτόματα υιοθετήθηκε τη νύχτα, Δευτέρα προς Τρίτη, όταν έληξε η προθεσμία και επειδή το Συμβούλιο δεν είχε εκφραστεί. Αυτή η μεταφορά, αυτό το έμβασμα λοιπόν ε, de facto εγκρίθηκε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα ενός ε, πιθανού διορθωτικού προϋπολογισμού στις αρχές του επόμενου έτους. Και ποιο θα ήταν το αδύναμο στοιχείο αυτού. Δεν μπορώ να σας πω καταρχήν από την άποψη της Κομισιόν εμείς φτιάχνουμε τον προπολογισμό με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας από τις γενικές ε, τεχνικές διευθύνσεις και από τα κράτη-μέλη. Και βεβαίως υπάρχουν αδύναμα σημεία, τα οποία θα μπορούσα να σας αναφέρω και να εντοπίσω και όπως και εσείς τα όσα περικόπησαν από το Συμβούλιο. Στο βαθμό που οι πιστώσει πληρωμών περικόπτονται σε σχέση με την πρόταση τη Κομισιόν, μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρχει μια αδυναμία σε εκείνο το σημείο, διότι ξεκινήσαμε από την υπόθεση ότι αυτές οι πιστώσεις πληρωμών θα χρησιμοποιούνταν. Αυτά μπορώ να πω, Πρόεδρε, σε σχέση με τα ερωτήματα που τέθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προτείνω τώρα να περάσουμε στις ψηφοφορίες και να ξεκινήσουμε από το 11, όπως μας ζήτησε ο εισηγητής, από το διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 5 και να ψηφίσουμε και τη νομική βάση και το διορθωτικό προϋπολογισμό, το συμπληρωματικό που είναι απαραίτητος για να χρηματοδοτηθούν οι σεισμοπαθείς στην ε, Εμιλία Ρωμάνα με ύψος 570 εκατομμύρια ευρώ. Ψηφίζουμε λοιπόν την έκθεση Φραντζέσκα Βαλτζάνη και Φερνάντες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δύο. Αποχές. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι σεισμοπαθείς θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Συγχαίρω τους ηγητές και χάρη στην αποφασιστικότητά τους καταφέραμε τουλάχιστον αυτό το θέμα να το διεκπαιρεώσουμε. Ε, υπάρχουν μεταφορές πιστώσεων στο σημείο 23, Φραντσέσκα. Θα μας τις παρουσιάσετε εντάχει, Φραντσέσκα. έχουμε μεταφορές πιστώσεων που σχετίζονται με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Μπορούμε να ψηφίσουμε κατευθείαν, γιατί ε, ε, δεν, υπάρχει δυνα... δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, συγγνώμη, δεν υπάρχει δυνατότητα ε, κινητοποίησης και πληρωμών, γιατί συνδέονται άμεσα με το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού περιθμών 6. Μα, μάλιστα, έχουμε όμως τρεις μεταφορές πιστώσεων, 36, 37 και 38. Είχαμε προβλέψει και τρεις ακόμη μεταφορές πιστώσεων, 36, 37 και 38. Θέλετε να τις, αναβάλουμε, καταρχήν μπορούμε να τις αναβάλουμε. Très bien. Donc, euh, sur ces virements, Madame le rapporteur. Η ρελτά η 37. Κοιτάξτε, 36, 37 και 38 στην πράξη δεν αφορούν το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, αλλά είναι εμβάσματα που αν δεν υπάρχει αντίρρηση μπορούμε να το ψηφίσουμε τώρα. Ωραία, ψηφίζουμε μαζί τι τρει μεταφορέ πιστώσεων. 36, 37, 38. Υπέρ. Κατά δύο κατά. Αποχές, μία αποχή. Κύριο Πάσκα. Εγκρίνονται λοιπόν οι τρεις μεταφορές πιστώσεων. Α, μπορώ να απελευθερώσω τους συζητητές, δεν τους διώχνω. Μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε τις ψηφοφορίες. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για έξι περίπου αιτήσει και εκθέσει που αφορούν την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, γιατί όπω μα ενημέρωσε η συγκήτρια, εφόσον δεν εγκρίναμε το διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 6, δεν μπορούμε να κινητοποιήσουμε το ταμείο αυτό. Οπότε θα ψηφίσουμε το σημείο 20, την γνωμοδότηση δηλαδή του κυρίου Σταυρακάκη, με θέμα τον Ενωσιακό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Έχετε τον κατάλογο ψηφοφορίας. Έκθεση στα βρακάκι. Έχετε όλοι τις ε, ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας, γιατί εγώ δεν την έχω. Voilà. <laughs> Bien. Alors, on va essayer de voter à main levée. Καλά, να ψηφίσουμε τότε διανατάσσεως της χειρός. Αλλιώς θα κάνω. Μπορούμε να ψηφίσουμε τις τροπολογίες 7 και 8 μαζί του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δύο κατά. Αποχές. Μία αποχή. Ωραία, εγκρίνονται. Τροπολογία 25 της Αντίνα Ιωάννα Βαλεάν. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος τέλος ψηφοφορίας 13 υπέρ 14 κατά και εγώ κατά ψηφίζω ούτως ή άλλως και χωρίς εμένα η πλειοψηφία είναι κατά Και άλλοι ξέχασαν τις κάρτες, μου όπως και εγώ, τις κάρτες τους όπως κι εγώ. Έχετε κάρτα κύριε Κλούτε. Έληξε ψηφοφόρια. Είστε κατά. <laughs> Εντάξει, εμείς αλληλοεξουδετερωνόμαστε. Εσείς υπέρ, εγώ κατά, σαν να μην υπάρχουμε. Α, είστε κατά κι εσείς. Α, τότε εντάξει, τότε συμπληρωνόμαστε. 13 υπέρ, 15 κατά, απορρίπτεται. Η τροπολογία 25. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 9 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Δύο αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Συμβατή της κυρίας Βαλεάν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27 Βαλεάν. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ε, Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 27. Μόνο εγώ δεν έχω την κάρτα μου, γιατί ο κύριος Κλούτη τη δικιά του τη βρήκε. Αποτέλεσμα. Τέλος ψηφοφορίας. Τι γίνεται, δεν ξέρει μαθηματικά ο υπολογιστής. 15 υπέρ 13 κατά συνένας εγκρίνεται η τροπολογία. Το 10 και 11 μαζί, ποιος είναι υπέρ. Κατά. 4 κατά. Αποχές εγκρίνονται. 28 βαλεάν. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ένας. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 και 13 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. 2. Αποχές. Εγκρίνεται με την ίδια διαφορά. 29. Βαλεάν. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 14 και 15 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δύο αποχές εγκρίνονται. 30 βαλεάν. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 αποσύρεται. Έχει αποσυρθεί. Τροπολογία, τροπολογίες 16 και 17 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Για τις αιτιολογικές σκέψεις τώρα έχουμε τις τροπολογίες 3, 4, 5 και 6 του συγγητού μαζί. Μπορούμε? Όχι, κάποιος δεν θέλει. Ποιος είναι υπέρ τη 3. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η γκου επέχει. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές και πάλι αποχή της Γκουε. εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά Αρτόγκ. Αποχές, χωρίς αποχές και αυτή εγκρίνεται με διαφορετικές πλειοψηφίες κάθε φορά όμως. Τροπολογία 19, Φερνάντες, ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 και 21 του κυρίου Κάζα. Μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 22. Φερνάντες. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 και 24. Το κύριο Κάζο. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, τροπολογία 1 και 2 του εισηγητού, μαζί, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δύο κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 18 του κ. Φερνάντες. Ο εισηγητή είναι υπέρ. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονικό τρόπο παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορίας. Ψήφισαν 26 υπέρ και εγώ 27, Δύο κατά και καμία αποχή. Εγκρίνεται συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Περνάμε τώρα στο σημείο 21. Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη της Μπάρβαρα Ματέρα. Έχετε το κατάλογο ψηφοφορίας. Αρχίζουμε. Τροπολογία 7 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 του κυρίου Γκάιερ. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Οπότε θα πρέπει να ψηφίσουμε όλες τις υπόλοιπες ψηφο, ε, τροπολογίες. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. 8 έως 14 της εισηγήτριας. Μέχρι τη 13. 8 με 13. από την 8 στη 13 μαζί. Γίνεται? Όχι. Αν υπάρχει συμμαχία Κορσικής Πορτογαλίας για να μας τη σπάσουν, εντάξει, ξεχωριστά. 8. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. 5. Κα... Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά 4 αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με μικρότερη διαφορά, αλλά όντω έπρεπε να τι ψηφίσουμε χωριστά. Ήταν διαφορετικό ο σχετισμό κάθε φορά. Η 15 αποσύρεται, 16 και 17 τη ηγήτρια. Μπορούμε μαζί. Όχι. 16. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πολύ διασκεδαστικό. Μια έχουμε πλειοψηφία της αριστεράς, μια πλειοψηφία της δεξιάς. 18 τώρα. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα ε, with the meaning in terms of. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, το πρόγραμμα παρτίζεται από μέχρι το Media Strand. Υπέρ εισηγήτρια, ποιος είναι υπέρ. Όλο το ΕΛΚ υπέρ, κατά. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κατά. Απόχες. Ε, το ΕΛΚ. Δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. 25 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 19. Ποιος είναι υπέρ της εισηγήτριας. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Για τις αιτιολογικές σκέψει τώρα. Τροπολογία 20. Κάζα υπέρ είναι η εισηγήτρια. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 της εισηγήτριας. ποιο είναι υπέρ. Κατά. 4. Η φιλελεύθερη είναι κατά. αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 21 Το κύριο Κάζα. Η είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για την 22 η συγκήτρια ζήτησε ψηφοφορία κατά τμήματα. Είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, το in από το in order του μέχρι το growth. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, investment centric knowledge. Γι' αυτό είναι κατά η συγκήτρια, υπέρ. Ο Γιάνν Μούλτερ κατά. Ο Γιάνν Μούλτερ πάλι και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια, αποχές είναι τραμερή εξήτηση της, Ολλανδική, της Ολλανδικής ψήφου. Δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Τροπολογία 4 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Τη εισηγήτρια μάλλον. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 του κυρίου Γκάιερ. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. 5 κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. 5 και 6 τη ηγήτριας. Μπορούμε να τι ψηφίσουμε από κοινού. Ναι. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. 3. Αποχέ Εγκρίνονται. Για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Να ψηφίσουμε μαζί τι τροπολογίε 1 και 2 της ηγήτριας. Υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. 2. απόχέ. εγκρίνονται Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, ψήφισαν όλοι, 22-23 και εγώ, δύο κατά και τρεις απόχες. Συγχαρητήρια στην καταπληκτική μας εισηγήτρια. Και περνάμε στην επόμενη έκθεση της ίδιας συζητητής, κυρίας Ματέρα, στο πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες. Μπορούμε τις δύο πρώτες τροπολογίες, την 6 και την 7, να ψηφίσουμε μαζί. Ποιος είναι υπέρ? Όχι. Δεν γίνεται. Την 6 ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. 2. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Η Θελελεύθερη και ο κύριος Χάρτονγκ. Εγκρίνεται διαφορετική πλειοψηφία μας. Η 8 αποσύρεται 12. Γκάιερ. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. 2. Αποχές εγκρίνεται. 9 και 10 μαζί γίνεται. Μα καλά επίτηδε το κάνετε για να με εκνευρίσετε. 9. Ε, ναι, Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 της συγκήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όντως. Ομολογώ ότι έπρεπε να ψηφίσουμε ξεχωριστά. Για τις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 3 της συγκήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 το κύριο Γκάιερ, Ποιο είναι υπέρ, κατά, 2 κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 4 αποσύρεται, 5 της ηγετίας, Ποιο είναι υπέρ, κατά, μία ψηφο. κατά, αποχέ εγκρίνεται. Για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματο. Τροπολογίε 1 και 2 μαζί, Ποιο είναι υπέρ, κατά, δύο κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Α, όχι. Ψήφισαν 25, συν 26, μήπως και κάποιος άλλος δεν πρόλαβε να ψηφίσει. Ένα μηχάνημα που δεν λειτουργεί. Τι είστε, υπέρ ή κατά. Υπέρ. Ωραία, 27 υπέρ. 2 κατά. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια και πάλι στην εισηγητριά μας. Euh, λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στις μεταφορές του ε, το προπολογισμό 2012 του κ. Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με αυτές τις προτάσεις ε, ε, τροποποίησης δεν υπάρχει πρόβλημα και όσον αφορά την πρόταση Μιλάμε για 5.000 ευρώ μόνο από την Επιτροπή των Περιφερειών που πρόκειται για δικαστικά έξοδα και δαπάνες σχετικές. Για την υπαριθμό 10 ε, ισχύουν αυτά που λέει στο Κόμπου News. Πρόκειται για 12.000 και όχι για 129.500. Και αυτή η μεταφορά, αυτή μάλλον η τροποποίηση, έχει να κάνει με την κινητικότητα και τις μεταφορές. 12.000 ευρώ, όχι 129. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, για την έγκριση αυτού. Σε σχέση με τις άλλες μεταφορές επιστώσεων και σε σχέση μάλιστα με αυτές που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να θυμίσω ότι αυτή η Επιτροπή επέβαλε μείωση 5% για τα ταξίδια. Αυτό, αυτή ήταν η συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις στην ομάδα εργασίας που υπάρχει σε αυτή την Επιτροπή και το Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Και ξέρω ότι η ομάδα εργασίας διαρκώς ενημέρωνε τους συντονιστές για τις ε, λύσεις που βρέθηκαν για αυτή τη μείωση του 5% στις ε, δαπάνες κάθε είδους ταξιδιού. Έτσι λοιπόν έγινε μια, με, βάση το ψήφισμα του Οκτωβρίου 2011. Έχουμε βάλει 10% στο αποθεματικό μέχρι ότου να οριστικοποιηθεί η απόφαση για το ταξίδι. Και αυτό το πετύχαμε μετά από τη δουλειά που έκανε η ομάδα εργασίας σε συνεργασία με το Προεδρείο. Και Άρα τώρα πρέπει να απελευθερώσουμε αυτό το απόθεμα. Τώρα, όσον αφορά την ε, ιστορία που είναι αρκετά γνωστή και για την οποία η Επιτροπή μας έχει δεσμεύσει εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα το ίδιο το Κοινοβούλιο, υποβλήθηκε ένα σχέδιο ένα business plan για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική και όλοι οι όροι που είχαμε επιβάλει για το αποθυματικό συμπεριλαμβάνονται εδώ. Άρα λοιπόν και αυτή η πρόταση τροποποίησης του προϋπολογισμού, αυτό το έμβασμα αριθμών 08 για την απελευθέρωση των 2 εκατομμυρίων που βρίσκονταν σε αποθυματικό και αυτό ότι ε, είμαι ε, θετικός. Είμαι λοιπόν θετικός υπέρ όλων αυτών των ε, μεταφορών πιστώσεων. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε πρώτα για τις μεταφορές της Επιτροπής των Περιφερειών, την 9 και τη 10. Ποιοι είναι υπέρ. Σας ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τώρα, για το Κοινοβούλιο. Η μεταφορά σε 07 υπέρ ποιοι είναι, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σε 08. Α, με συγχωρείτε, μία αποχή, μάλιστα. Σε 08. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Κύριε Κλούτε, υπέρ κατά είστε. Μάλιστα. Εποχέ εγκρίνεται με μια εποχή Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα, μάλλον σας προτείνω τώρα, νομίζω ότι ο κ. Αλφονσί βιάζεται. Γι' αυτό σας προτείνω να περάσουμε στο θέμα του κ. Αλφονσί που είναι το υπερθμό 9. Και είναι η έκθεση για την αλληλεία. Συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που ανακατεύετε την ημερήσια διάταξη, γιατί είναι τέτοιε υποχρεώσει μα. Πρόκειται για τη γνωμοδότησή μα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλασσίων Υποθέσεων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε την βιώσιμη αλληλεία και υδατοκαλλιέργεια και ανάπτυξη ισορροπημένης, ισορροπημένων δραστηριοτήτων, κυρίως στις παράκτητες περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την έντονη εντατική αλληλεία. Οι πυλώνες αυτής της πολιτικής βασίζονται σε μια πράσινη και ευφυή αλληλεία, υδατοκαλλιέργεια οικολογικής φύσης, αλληλεγγύη με τις περιφερειές και ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αυτό το, αυτή η, η πολιτική αλληλείας θα πρέπει να στηρίξει τη βιώσιμη αλληλεία γιατί όπως και όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα της αλληλείας είναι πως ακόμα δεν έχει βρει την ισορροπία της με τους πραγματικούς πόρους του φυσικού περιβάλλοντος και για να προχωρήσουμε προς καλύτερη απόδοση και καλύτερη ε, μετάλλευση των πόρων συμβατή με το περιβάλλον η Κομισιόν προτείνει να τονιστούν δύο μεγάλα μέτρα καταρχήν η κατάργηση των απορρίψεων και η μείωση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον μέσω πρακτικών αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας που με θετική ε, επιρροή στο περιβάλλον καθώς και το συντονισμό των θαλασσίων πολιτικών. Η βιώσιμη λοιπόν ανάπτυξη πρέπει να γίνει σύμφωνα με την Κομισιόν ενισχύοντα ε, την ε, εμπλοκή των ε, τοπικών φορέων. Επίση, είναι ενδιαφέρον ότι η αλληλευτική πολιτική για πρώτη φορά ενσωματώνει το ρόλο των γυναικών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση των επιχειρήσεων τη δίκηση των επιχειρήσεων και επίσης το πρόγραμμα αυτό προβλέπει να ευνοηθούν και αναβιώμενες δραστηριότητες που μπορεί να έρθουν και να συμπληρώσουν τα έσοδα των αλλιών που σήμερα πολύ δύσκολα τα βγάζουν πέρα μόνο και μόνο από την αλλία. Για μας πρόκειται για προσανατολισμούς λοιπόν ενδιαφέροντες. Υπάρχουν και άλλοι προσανατολισμοί που νομίζουμε ότι πρέπει να υποστηριχτούν και είναι η αύξηση του κονδυλίου για τη σύλλογη των στοιχείων και για τη τις πιο εμπεριστατωμένες επιστημονικές απόψεις που δεν θα δώσουν λαβή για πολεμικές όπως τις γνωρίζουμε πολύ συχνά ανάμεσα στους επαγγελματίες και τους ακαδημαϊκούς για τον καθαρισμό των ποσοστώσεων και των ορίων της αλληλευτικής προσπάθειας σε σχέση με τα διάφορα είδη και τις διάφορες θαλάσσιες λεκάνες. Στη συνέχεια, για να αντιμετωπιστούν, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η Κομισιόν προτείνει προγραμματισμό 2014 με 20 με αύξηση 2,7% των ποσών σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, πράγμα που θα πρέπει να επιτρέψει να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι υποχρεώσεις, να καλυφθούν μάλλον όλες αυτές οι υποχρεώσεις. Υπάρχουν τώρα κάποιες τροποποιήσεις, ορισμένοι θα έλεγα Ορισμένε τροποποιήσει είναι κοινέ με τα όσα κάναμε για άλλα ταμεία. Όλε αυτέ οι προτάσει και οι άξονε δαπανών ισχύουν μόνο αν τα κράτη δεχτούν να δώσουν του απαραίτητου πόρου στη μελλοντικό PDP. Και άρα προφανώ, αν υπάρξουν περικοπέ, θα πρέπει να μπορέσει το Συμβούλιο να πει ακριβώ πού θα πρέπει να γίνουν αυτέ οι περικοπέ. Δεύτερος στόχος που έχουμε για το σύνολο των κονδυλίων είναι να διατηρηθεί η διοργανική συμφωνία που αναθέτει συγκεκριμένο ρόλο στο Ευρωκοινοβούλιο και έπειτα συγκεκριμένα μέτρα για συγκεκριμένα προγράμματα προτείνουμε μέσω τροπολογιών ε, δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι να λάβουμε υπόψη τη σημασία και το ρόλο της παράκτιας αλληλείας για την χωροταξία του παράκτου περιβάλλοντος και έτσι ώστε για να μην συμβεί δηλαδή πάλι όπως σε προηγούμενες περιόδους να μην αποτελέσει το αδύναμο κρίκο αυτού του κλάδου που βρίσκεται εκτεθειμένος στην μείωση ε, της δραστηριότητα, γιατί εδώ έχουμε φτάσει σε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή των παρακτήων περιοχών. Και δεύτερος προσανατολισμός, δεύτερη κατεύθυνση είναι να θυμίσουμε ότι υπάρχουν παραδοσιακές οργανώσεις, κυρίως στον μεσογειακό χώρο, αλλά φαντάζομαι ότι και αλλού υπάρχουν οργανώσεις που συντονίζουν και που οδηγούν ώστε οι επαγγελματίε και οι ασχολούμενοι στην αλληλεία ε, με βάση ε, αρχαία... Ε, αρχαίγονες μεθόδους ε, ε, πολύ παλιές να συνεχίσουν, να μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν αυτές τις δραστηριότητες με βάση την κοινή πολιτική ε, αλληλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά εν ολίγης, αυτά που λέει αυτή, η γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Όντως, σε θέματα αλληλείας η Μεσόγειος από την αρχαιότητα έχει ένα σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης ε, πολύ ιδιαίτερο που αποδείχθηκε και πολύ αποτελεσματικό άλλωστε τουλάχιστον σε ό,τι φορά τις νότιες, τη, νότια, τη βόρεια συγγνώμη, όχθη της Μεσογείου. Ε, σχόλια δεν έχετε, έτσι. Θυμίζω ότι για την έκθεση Αλφόνση η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών εκπνέει αύριο στις 10. Θα ψηφίσουμε στις 6 Δεκεμβρίου για να μπορέσει στις 19 Φεβρουαρίου να ψηφίσει η Επιτροπή Αλίας. Άνετες είναι οι προθεσμίες για να φτάσει στην Ολομέλεια το Μάρτιο η έκθεση. Λοιπόν, σλάλομ κάνω εδώ πέρα με την ημέρηση διάταξη για να προσπαθήσω να βολέψω όλους σας. Είναι λίγο περίπλοκα αυτά Τώρα γυρνάμε λίγο πίσω, στο σημείο 25, διότι πρέπει να φύγει η κυρία Μόνικα Χολμάγερ. Αν μπορεί να παραμείνει λίγο ο κύριος Γενικός, αμέσως μετά θα πάμε στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συγγνώμη που σας καθυστερώ. Αλλά είναι λίγο περίπλοκη σήμερα η συνεδρίαση. Αγαπητή Μόνικα, πολιτική ακινήτων, τι νέα έχουμε. Ε, πάρα πολύ σύντομα θα σας τα πω. Ε, σε συμφωνία με τους συναδέλφους, ε, σήμερα δεν θα κάνουμε μεγάλη συζήτηση. Μια γνωμοδότηση θα καταθέσουμε στις 3 Δεκεμβρίου, γιατί παραμένουν ακόμα κάποια ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γι' αυτό δεν μπορούμε σήμερα να συνεχίσουμε μια συζήτηση όπου δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα. Είναι πολύ μεγάλο το έργο και κανονικά είναι σωστός ο προγραμματισμός με σύνεση, είναι νωρίς ακόμα. Περιμένετε, θα σας φέρουμε μια συγκεκριμένη γνωμοδότηση για να έχουν απαντηθεί κάποια θέματα. 10% αποθεματικό και κάποια τέτοια πρέπει να κλειδώσουν για να μην ε, εκραγεί το κόστος. Ωραία. Μα λέγει λοιπόν η συγκήτρια ότι σήμερα δεν είναι σε θέση να μα παρουσιάσει το θέμα, διότι δεν έχουμε όλε τι απαραίτητε πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε σα προτείνω να το αναβάλουμε αυτό το θέμα και τη συζήτηση και την ψηφοφορία για την επόμενη φορά, την ενδεχόμενη ψηφοφορία χρειαστεί όταν θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Et donc, euh, donc Α, γνωμοδότησα κάνουμε. Ναι, ναι, εντάξει. Συμφωνούμε να γνωμοδοτήσουμε. Συζήτηση θα γίνει. Και ψηφοφορία για το περιεχόμενο της γνωμοδότησης. Ωραία, σας ευχαριστώ. Και τώρα, επανερχόμαστε στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνοψίζω. Σε μία φράση, πώς έχει η κατάσταση. Η Κυπριακή Προεδρία τελικά κατέθεσε ποσά λεγόμενα συμβιβαστικά εξ ονόματος Κυπριακής Προεδρίας για να ε, ολοκληρωθεί το πακέτο ε, της διαπραγμάτευσης και μετά από λίγες μέρες, χτες συγκεκριμένα, στις 12 και 10 το βράδυ, Ο πρόεδρος να πάει, ξέρετε, είναι νικτόβιο on. Δηλαδή βασικά 24 ώρες, 24 ώρες εργάζεται ο άνθρωπος. Ε, εξέδωσε τα δικά του ποσά που διαφέρουν αισθητά από τις συμβιβαστικές λεγόμενες προτάσεις της Κυπριακής Προεδρίας. και θα τα υποβάλει αυτά ε, τα ποσά στις 22 και 23 Νοεμβρίου στο Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πριν δώσω το λόγο στους παρόντες εισηγητές, η Βάιλο, συμφωνείς να ακούσουμε πρώτα το Γενικό Διευθυντή. Τι να, τι να πω, λέει ο κύριος Κάλφιν. Ε, ακούσουμε τον κύριο Γενικό πρώτα. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί να γίνει μακρά συζήτηση στο ΚΟΡΕΠΕΡ, στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, επί της πρότασης του ε, Πρόεδρου Βαν Ρομπάη και μίλησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας πω τι είπε στο ΚΟΡΕΠΕΡ η Κομισιόν σήμερα. Πρώτον, ότι θεωρεί ότι η πρότασή της ήταν η πιο ισόρροπη. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή. Και εξέφρασε τη λύπη της για τις επιπλέον περικοπές που προτείνονται. Ε, δεύτερον, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αναγνώριζε το γεγονός ότι η πρόταση του κύριου Φανοπάη σέβεται την ισορροπία που είχε προτείνει στην αρχική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και στα πλαίσια του προηγουμένου σχολείου μου, αυτό είναι κάτι το θετικό. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της, διότι ε, στους ιδίους πόρους έγιναν πρόοδοι, με τριοπαθείς μεν σε ό,τι αφορά το φόρο θέμενης αξίας, αλλά με στόχο για το 2021 παρόλα αυτά. Δηλαδή να έχουμε το νέο ΦΠΑ τότε και το φόρο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ακόμα και υπό μορφή ε, ενισχυμένης συνεργασίας, τελικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ίδιος πόρος για να χρησιμοποιηθεί και στον οποίο θα μπορούσαν να καταφεύγουν τα κράτη-μέλη που θα τον επιβάλλουν στην επικράτειά τους. Τελευταίο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διατράνωσε την υποστήριξη της προς τον κύριο Φανρόμπα στη διαδικασία αυτή. Αυτά ήταν τα τέσσερα σημεία που είχα να σας αναφέρω για να σας ε, δείξω πού προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 75 δισεκατομμύρια είναι οι περικοπές και γίνονται 80 αν ε, βάλουμε και τα ποσά εκτός του πλαισίου των πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριο Χάρτονγκ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα είμαι ευγνώμων για την καθημερινή δουλειά τη Κυπριακή Προεδρία, μάλλον την ημερήσια δουλειά τη προεδρία και την νυχτερινή δουλειά του κυρίου Φον Ρομπάη. Είμαι πολύ, περίεργη, ε, ε, πολύ περίεργος να δω τι θα βγει τελικά από το Συμβούλιο, αφού δουλεύουν τη μέρα η Κυπριακή Προεδρία και το βράδυ τη νύχτα ο κύριος Πανρόμπα. Ευχαριστώ. Θα διαπιστώσετε κύριε Χάρτονγκ ότι οι δύο προτάσεις, η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας και η πρόταση Βαν Ρομπόη διαφέρουν. Το συνολικό ποσό, ως προς το συνολικό ποσό, αλλά κυρίως ως προς την κατανομή. Η Έχετε κάποιο σχόλιο. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο κύριε Πρόεδρε. Ευθυγραμμιζόμαστε με τη θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευελπιστούμε ότι θα εμείνει στη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι την επίτευξη συμφωνίας. Σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση έκθεση και με βάση αυτή που εγκρίναμε με μεγάλη πλειοψηφία, δεν μπορούμε να δεχτούμε προτάσεις τέτοιων περικοπών του προϋπολογισμού, ούτε ε, περικοπές χωρίς αναθεώρηση σημαντικών πολιτικών. Και δεν ε, υπάρχει αρκετή ελαστικότητα στην πρόταση. Ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις ε, για συμφωνία στους ιδίους πόρους. Το μόνο θετικό που έχει πρόταση σε σχέση με τις μέχρι τώρα υποβληθήσεις είναι η ετοιμότητα για διάμεση αναθεώρηση. Έχουμε τώρα διοργανική συμφωνία μέχρι στιγμής, αλλά με, ανέκαθεν παρακόλληλε τη διαδικασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς επιμένουμε στην διάμεση αναθεώρηση και θέλουμε να είναι δεσμευτική αυτή τη φορά και να συνδέεται με τον προϋπολογισμό του 2018 που βρίσκεται στα μέσα της περίοδου των ε, δημοσιονομικών προοπτικών. Αυτό είναι το μόνο θετικό στοιχείο, γιατί όλα τα υπόλοιπα σημεία που είναι πολύ σημαντικά για το Κοινοβούλιο δυστυχώ δεν μα ικανοποιούν, ε, γιατί η τελευταία πρόταση παλιδρομεί σε σχέση με τι προηγούμενε. Ευχαριστώ, Ιβάιλο. Ιαν Ευχαριστώ. Η Επιτροπή μα είπε ότι υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία για του ίδιου πόρου. και περιμένουμε με ενδιαφέρον ε, τις αντιδράσεις ε, στο Συμβούλιο των κρατών μελών. Το σύστημα για την ίσπραξη παραδοσιακών ιδιοπόρων όπως ε, των τελωνιακών δεσμών, αυτό το σύστημα παραμένει αμετάβλητο, αλλά τροποποιούνται τα ποσά που μπορούν να κρατήσουν τα κράτη-μέλη από 25 το ποσοστό κατεβαίνει στο 15%. Δεν νομίζω να ικανοποιήθηκε πολύ με τις αλλαγές αυτές ο κύριος Χάρτονγκ. Επίσης, βλέπετε περικοπές, μερικές από τις επιστροφές. Ο Βαν προτείνει εφάπαξη για τη Γερμανία, τις κατοχώρες και τη Σουηδία. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κρατά την αιώνια αυτή επιστροφή, το αιώνιο αυτό δικαίωμα επιστροφή στο rebate που έχει και όλες οι διορθώσεις θα χρηματοδοτηθούν πλήρως από όλα τα κράτη-μέλη με βάση την κλίδα του ΑΕΠ. Κάτι που είναι θετικό για τη Δανία, γιατί πληρώνει πολλά για τη Βρετανική επιστροφή. Γι' αυτό ζητήσαμε και εμείς για μας επιστροφή. Αλλά βέβαια άλλο είναι το σκεπτικό. Και δεν είναι και εύκολο να πάρει η Δανία rebate επιστροφή. Τώρα για τους ίδιους πόρους αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε στη βάση του ΦΠΑ που είναι πιο γνωσ... ο πιο γνωστός ίδιος πόρος. Χαίρομαι που αναφέρεται αυτό και ότι ο νέος πόρος ΦΠΑ θα πρέπει να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα από την 1η Πρώτου 2021. Μιλάμε για απότερο μέλλον. Ε, τις επόμενες δηλαδή δημοσιονομικές προοπτικές, στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο κύριος Ζωνζόν είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με ενισχυμένη συνεργασία να χρησιμοποιηθεί για τα δύο τρίτα των εσόδων, ώστε να μειωθεί αντίστοιχα η εθνική εισφορά. Φαίνεται ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη κάποιες προτάσεις του Κοινοβουλίου δεν αναφέρονται τα έξι σημεία του δικού μας ψηφίσματος παρόλο που κατά τη γνώμη μας ήταν πολύ θετικά και θα διευκόλυνε και το Συμβούλιο αλλά ε, επαναλαμβάνω περιμένουμε με ενδιαφέρον την αντίδραση του Συμβουλίου. γιατί θεωρώ ότι πολλά κρατημέλη θα δυσανασχετήσουν με την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ, Αν. Όπως είπαν και η Αν και ο κύριος Ζων ε, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τους ίδιους πόρους, η πρόταση δεν είναι ιδεώδης, αλλά αυτό που έχει προτείνει μέχρι τώρα ο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι μια σοβαρή αν άλλο βάση και χαίρομαι προσωπικά γιατί είναι ένα θέμα που και προσωπικά ο πρόεδρος Βαν Ρόμποϊ ε, ε, υπέβαλε και μάλιστα τροποποίησε τη δική του θέση λαμβάνοντας υπόψη τα δικά μας σχόλια. Και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποστήριξε τη θέση αυτή και απέναντι στον πρόεδρο Βανεροπόη. Τώρα, για τη συνέχεια. Καταρχήν, να λάβουμε υπόψη ότι ολοκληρώνεται όλη η προπαρασκευαστική φάση των διαπραγματεύσεων που ουσιαστικά τώρα ξεκινούν στο Συμβούλιο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα συνεχιστούν με τη διαδικασία της σύμφωνης γνώμης μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου μετά τη διάσκεψη κορυφής. Καταφέραμε οι προεδρίες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους τις δεσμεύσεις που είχε λάβει η Ουγγρική Προεδρία απέναντι στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή να αναμειχθεί το Κοινοβούλιο, να εμπλακεί από την πρώτη μέρα στις ε, προπαρασκευαστικές συζητήσεις και στην προετοιμασία ακόμη των διαπραγματεύσεων που γίνονται στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Δεν σημείωσα λεπτομεριακά όλε τι συνεδριάσει. Μία το μήνα κατά κανόνα γινόταν και σε όλε συμμετείχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Προσκληθήκαμε σε όλες τις άτυπες ε, συνεδριάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Μία φορά από την Δανική Προεδρία και δύο φορές από την Κυπριακή Προεδρία. Έτσι μπορέσαμε μη τι άλλο να συμμετέχουμε στις συζητήσεις. Ε, δώσαμε το παρόν και παρουσιάσαμε την ε, άποψή μας και μάλιστα ελήφθη υπόψη και η δική μας θέση μαζί με τις άλλες. Έτσι δημιουργήσαμε και κάποιες οικειότητες και κάποιες συμμαχίες για ορισμένα θέματα. Με κάποιες κυβερνήσεις και για άλλα θέματα με άλλες κυβερνήσεις. Και με προσωπική πρωτοβουλία του Πρόεδρου Σούλτς, η ομάδα των φίλων της συνοχής συνεδρίασε προχθές στους χώρους, στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάλεσε τον πρόεδρο Σούλτς και τον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών σε ένα τμήμα τουλάχιστον των, της συνεδρίασης. Και εκεί ο πρόεδρος Σούλτς παρουσίασε τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα στα σημεία εκείνα που ευθυγραμμίζονταν με τις ε, θέσεις των φίλων της συνοχής. Γιατί ούτε και οι 15 χώρες ε, της ομάδας των φίλων της συνοχής συμφωνούν ε, εφόλης της ύλης θέλουν ένα υψηλό προϋπολογισμό, ειδικά για την πολιτική της συνοχής, ένα παχυλό προϋπολογισμό, αλλά για παράδειγμα για τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα που θα πρέπει να συνοδεύει κάποιες ενισχύσεις, είναι το αντιστάθμισμα κάποιων ενισχύσεων, γι' αυτό δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των 15 χωρών των φίλων της συνοχής. Επίσης, για τη χρηματοδότηση του μηχανισμού συνδέοντας την Ευρώπη και για το κατά πόσο ένα τμήμα της χρηματοδότησης ε, θα πρέπει να προέλθει από την πολιτική της συνοχής, από τον προϋπολογισμό της συνοχής. Ούτε και εκεί συμφωνούν όλες οι χώρες των φίλων της συνοχής. Πάντως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συνεχείς επαφές και με τις 27 χώρες εδώ και ένα χρόνο περίπου. Αλλά αυτή η προπαρασκευαστική φτάση, ε, φάση φτάνει στο τέλος της. Η Κυπριακή Προεδρία έδωσε αντίγραφο τις θέσεις των στον πρόεδρο Βαν και από τις 5 Νοεμβρίου ο πρόεδρος Βαν ξεκίνησε τις διμερείς διαπραγματεύσεις. της ε, εξομολογείς όπως λέμε στην ε, κοινοτική αργό. Οπότε κάθε αντιπροσωπεία έπρεπε να πάει για εξομολόγηση και πήγαμε και εμείς, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να εξομολογηθούμε στον ε, επικεφαλής του γραφείου του Πρόεδρου Βαν Ρομπόη. Και μετά από εκτενή και βρυθή συζήτηση, παρουσία της κυρίας Καντρίντε, που εκπροσωπούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εξομολογητήριο, παρουσίασε, παρουσιάσαμε τις θέσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημειώθηκαν οι απόψεις μας και τώρα να πω και στον πρώτο Βαν Ρομπόη να αντιλήσει κάποια συμπεράσματα. Γιατί αυτός ε, χειρίζεται αυτές τις διαπραγματεύσεις. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα. Την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε την τελευταία ε, σύσκεψη με το τρίο των Προεδριών με τη μορφή ε, γεύματο εργασία. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα στις Βρυξέλλε, ενώ όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα μεταβούν στο, Στρα... Στρασβούργο, ή θα είναι στο δρόμο προ το Στρασβούργο. Και όλη η αντιπροσωπεία μα είναι προσκεκλημένη στο γεύμα αυτό εργασία. προκειμένου να ετοιμάσουμε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που θα λάβει χώρα την Τρίτη στις Βρυξέλλες. Στο μεταξύ όλοι θα έχουμε πάει στο Στρασβούργο βέβαια και θα είναι ευκαιρία για τους ε, Υπουργούς ε, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ε, να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων για τις προτάσεις Βαν Ρομπόη. Τώρα, το πακέτο το υποδιαπραγμάτευση είναι πλήρες, γιατί περιλαμβάνει και συγκεκριμένα ποσά, οπότε δεν θα το τροποποιήσει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Αυτό που θα δοθεί στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τις επόμενες εβδομάδες είναι το σχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ετοιμάζει ο πρόεδρος Βαν Ρομπόη. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων γενικώ δεν θεωρείται αρμόδιο για να τροποποιήσει το σχέδιο συμπερασμάτων του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά θα το συζητήσει και ο καθένα θα δώσει τι απόψει του, μετά ο πρόεδρος του Συμβουλίου να τροποποιήσει ενδεχομένω τα συμπεράσματα ανάλογα με τη συζήτηση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Κατόπιν, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την ε, προπαρασκευαστική και πάλι φάση σταματάει εδώ. Στην ομάδα επαφή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, προβληματιστήκαμε και το συζητήσαμε και με τον πρόεδρο Σούλτς για το κατά πόσο το Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει και θα συνεχίσει τέτοιου είδους επαφές και σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπως είχαμε μέχρι τώρα με το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και κρίναμε ότι δεν είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο. Ότι δεν συνάδει με το πνεύμα της συνθήκης αλλά ούτε και με το γράμμα της συνθήκης. Κρίμα, αλλά έτσι έτσι έχουν τα πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε και το γράμμα και το πνεύμα της συνθήκης. Άρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα γίνει κανονικά με βάση τη διαδικασία. Θα προσκλήθει φυσικά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αρχική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θυμοτυπικά κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ξεκινά με μία ανακοίνωση του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενημερώνει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε στην Ολομέλεια είτε στις αρμόδιες επιτροπές ανάλογα με τη διαδικασία που ισχύει για τα διάφορα θέματα και για τα θέματα που αφορούν φυσικά την ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Βέβαια, ένα θα είναι μόνο το θέμα τη ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου, το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και ο πρόεδρο Σούλτ με βάση το ψήφισμα που εγκρίναμε, θα υπενθυμίσει στο Συμβούλιο της θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέχασα να σας πω ότι αναφέραμε το θέμα, ερωτήσαμε μάλλον, αν θα έπρεπε να υιοθετήσουμε ένα τελευταίο ψήφισμα την παραμονή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είχαμε διατηρήσει αυτή τη δυνατότητα. Τελικά όμως δεν θεωρήσαμε πως είναι απαραίτητο αυτό γιατί το ψήφισμα που υιοθετήσαμε τον περασμένο μήνα ήταν πολύ καλό. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, σχεδόν 80% των ψηφισάντων. Και εξάλλου, για τα νούμερα που έχουμε επιτάπει οι συγκητέ έχουν αντιδράσει, οι πολιτικέ ομάδε έχουν αντιδράσει, οπότε δεν θεωρήσαν πω ήταν σκόπιμο να προχωρήσουμε σε καινούργια ψηφοφορία. Αντίθετα, βεβαίω, όπω κάνουμε πριν από κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα γίνει την Τετάρτη το πρωί μια μεγάλη συζήτηση που θα ξεκινήσει με δηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας και του Προέδρου της Κομισιόν για τα θέματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μετά έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος Σούλτς θα παρουσιάσει την πρόταση του Κοινοβουλίου. Ίσως να γίνει μια αρχή συζήτηση ή μια ανταλλαγή ερωτήσεων. Έπειτα θα αποσυρθεί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα γίνει χωρίς εμάς, ερήμην μας. Στη συνέχεια θα δούμε επί τη βάση των συμπερασμάτων πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία αν υπάρξει ομόφωνη ε, πρόταση, απόφαση μάλλον θα δούμε και οι συγητές θα μας κάνουν προτάσεις για το πώς θα προετοιμάσουμε τη δική μας αντίδραση και την ψήφα μας. Εάν κάτι που φαίνεται πιθανότερο δεν καταφτάσουν με την πρώτη σε πλήρη συμφωνία, τότε θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί κάλλιστα να βρεθούμε σε μια διάμεση κατάσταση, πράγμα που κατά τη γνώμη μου θα ήταν θετικό για όλους. Όπου δηλαδή μετά από πολύ μακρές και εις βάθος ανταλλαγές απόψεων που ο καθένας θα έχει διώσει την, την άποψή του και την άποψη της χώρας του, θα έχουν προχωρήσει για κάποια θέματα και αρχές. Θα έχουν προχωρήσει για να βάλουν τις βάσεις για έναν πρώτον τελικό συμβιβασμό. Και τότε μπορούμε βεβαίω να φανταστούμε ότι το Κοινοβούλιο θα αντιδράσει σε αυτή την πρώτη φάση διαπραγματεύσεων και ότι εν τέλει θα είναι μια δυνατότητα για το Κοινοβούλιο και ένα τρόπο για να ξεκινήσει μια μορφή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πράγμα που μπορεί και να διευκολύνει στη συνέχεια την επανέναρξη των εργασιών σε μια επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ούτω ώστε το Κοινοβούλιο και η άποψή του όντας γνωστή, να ληφθεί και υπόψη. τότε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα κινητοποιηθεί για να προετοιμάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το, θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε εμεί την θέση μας σε επίπεδο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Απτά. Σας ευχαριστώ και κλείνω τη συζήτηση. Ε, le MFF et euh, je reviens au point... Euh, και έρχομαι που ήταν ο εισηγητή, ποιο είδε κάποιο μήπω βιάζεται. Γιούτα λοιπόν, η Γιούτα βιάζεται. Είναι και αντιπρόεδρο, ήταν πολύ διακριτική αλλά πολύ προσεκτική εξ αρχή. και θέλησε λοιπόν τώρα να εξετάσουμε το 6, σημείο 6. Μάλιστα. Περί τίνο πρόκειται τώρα στο 6. Η τραπεζική αρχή. Ο ε, οργανισμός είναι, agency αυτός, που εμείς ε, καθιδρύσαμε μόλις πέρσι, αλλά με την ομοθεσία που τώρα πρόκειται να εγκριθεί εν ώψη της Τραπεζικής Ένωσης και εκεί ανήκει και η Τραπεζική Εποπτεία, θα πρέπει να το δούμε. Αυτά τα πράγματα είναι κυρίως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έπρεπε λίγο να προσαρμόσει τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, ΕΜΠΑ. Αυτό είναι λοιπόν το αντικείμενο. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της ΕΜΠΑ περιγράφονται στο κείμενο αυτό. Ενδεχομένως θα ε, αυξηθούν τα καθήκοντά της. Είμαστε μόλις στην αρχή της νομοθετικής διαδικασίας τονίζουμε επιμόνως, όπως πάντα, ότι ε, μαζί με το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 47 της Διοργανικής ε, Συμφωνίας μας, θα συζητήσουμε ε, και θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Πλην όμως, ταυτόχρονα λέγουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλουμε ένα νέο δημοσιονομικό δελτίο μόλις ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία. Στο παρελθόν είδαμε ξανά και ξανά ότι με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την ίδρυση του εκάστοτε οργανισμού δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε εάν κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας προστίθεντο στο παρελθόν και νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Αυτό ξεκίνησε από την ΕΣΜΑ για τη θάλασσα και τώρα κάθε φορά ζητάμε τροποποιημένο δημοσιονομικό δελτίο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είμαστε οπλισμένοι και κατοχυρωμένοι για το επόμενο βήμα, για την επόμενη διαδικασία, την ενιάψια του προπολογισμού. Να μην είμαστε συνεχώς τριμωγμένοι στη γωνία και να μην μας φτάνουν τα λεφτά. Η τρίτη τροπολογία αφορά το εξής. Περιμένουμε λοιπόν η ΕΜΠΑ να έχει επαρκή ε, σπόρους και οικονομικούς αλλά και ανθρώπινους, να στελεχωθεί καλά για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο της. Αυτό μάλλον έτοιμα είναι, δεν είναι τυπικά νομικά τροπολογία αυτή καθ' αυτή, αλλά νομίζω θα πρέπει να υποθεί επιγόντως. Και ελπίζω οι συνάδελφοι της Οικονομικής Επιτροπής να συμφωνήσουν με τις τροπολογίες μας και να τις συμπεριλάβουν τελικά στην έκθεσή τους και να μην μπορεί να γλιστρήσει το Συμβούλιο. Αυτά σύντομα και τα πιο σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ Γιώτα. Ιαν Γένσεν. Υποστηρίζω τη έκθεση της Γιώτα τη γνωμοδότηση μάλλον είναι σαφέστατη. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο και αυτές τις εποπτικές αρχές, τις τρεις ε, νέες δομές τους οργανισμούς που εν μέρη χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη και αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό συζητήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, την οποία συναντούν σε τακτά χρονικά διαστήματα και ε, διαμαρτύρονται και παραπονιούνται ότι τους δυσκολεύει πολύ η ζωή γιατί δεν έχουν ένα δημοσιονομικό κανονισμό να τηρήσουν, έχουν πολλούς. Και είναι βαριά η γραφειοκρατία και το διοικητικό άχθος. Τι ζητώ λοιπόν. Ναι, είναι ενταγμένη στον κοινοτικό προπολογισμό και σε μια μετάβαση που τελικά να χρηματοδοτούνται από τέλη ε, που καταβάλει ο ίδιος ο τομέας. Αυτό συμβαίνει σε κάποιες χώρες. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας ε, χρηματοδοτεί μερικός ή ολικός ε, τις αποπτικές του αρχές. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει εμεί ω Επιτροπή Προπολογισμών να προβληματιστούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Μπορούμε κάποια στιγμή να το συζητήσουμε και αυτό για την ένταξή του στον προπολογισμό, γιατί είναι πραγματική τους επιθυμία και θα τους διευκόλυνε πολύ τη ζωή, όσο και την αποτελεσματική του λειτουργία. κυρία Χάουκ, σε μια αιτιολογική σκέψη. Μπορούμε να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέω εγώ, να μας κάνει μια πρόταση. Πρέπει να αλλάξουν και οι βασικοί κανονισμοί, έτσι, ή ο βασικός κανονισμός. Και μπορούμε να το ζητήσουμε αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια αιτιολογική σκέψη. Πώς σας φαίνεται αυτό. Το κατανοώ. αυτή η χρηματοδότηση μισό-μισό ήταν ένα τέχνασμα, γιατί ο δικός μας τίτλος 1α είχε στερέψει από χρηματοδότηση. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσουμε, αν θα πετύχουμε κάτι ουσιαστικό έτσι, αλλά από την πρώτη πρώτου του 2014 είναι σαφές ότι πρέπει να μας προβληματίσει ξανά αυτό, γιατί πρέπει να αλλάξουμε τις κατηγορίες και τους τίτλους στον προπολογισμό. Όταν θα το καταθέσει η Κομισιόν βεβαίως μπορούμε και αυτό να το συμπεριλάβουμε. Ο Πρόεδρος, καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Όντω και τα πράγματα θα περιπλακούν ακόμη περισσότερο από την τεχνική και γραφειοκρατική άποψη με τη δημιουργία μια ενισχυμένη εποπτεία που ανατίθεται βασικά στην ΕΚΤ. Και άρα θα πρέπει αυτό να το παρακολουθούμε πολύ στενά. Ευχαριστώ, Γιούτα. Η υποβολή τροπολογιών 19 Νοεμβρίου το μεσημέρι στις 12. Θα ψηφίσουμε 3 Δεκεμβρίου ώστε η ΕΚΟΝ να μπορέσει να ψηφίσει το Μάρτιο. Και στη συνέχεια θα δούμε στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ και περνάμε στο σημείο 7. Ειδική έκθεση υπαριθμών 6 για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η κυρία Νέσκι, αγαπητή Ναντέζνα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θέλω να καταστήσω σαφές ότι εξαρτάζουμε ένα περιορισμένο φάσμα, δηλαδή με βάση την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για την αποτελεσματική εφαρμογή, εκτέλεση μάλλον, του εις βοήθειας προς την τουρκοκυπρική κοινότητα και όχι το κατά πόσο επιτεχάνει το στόχος της συμφιλίωσης ε, Πρόκειται για μια βοήθεια μέχρι την, την ολοκληρωμένη λύση στο Κυπριακό επετεύχθη για την περίοδο που ξεκινά το 2006 για προγράμματα που δίνονται όχι μόνο νέα, για προγράμματα όχι μόνο νέα αλλά και σε υφιστάμενα προγράμματα ε, για την εισαγωγή καταλήλων μηχανισμών εφαρμογής. Αυτό σημαίνει στήριξη για την επιτυχή χρηματοδότηση, μάλλον ε, ναι, εφαρμογή της χρηματοδότησης. Η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 16 Δεκεμβρίου στις 10 η ώρα και θα ψηφιστεί το Δεκέμβριο πριν την τελική ψηφοφορία που θα γίνει στην αρμόδια της Επιτροπή, την ΚΟΝΤ, την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Σας ευχαριστώ. Όντως πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα λοιπόν, το οποίο δεν μπορεί οριστικώς να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, διότι έχουμε προβλέψει ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Οπότε η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι αύριο μέχρι τις 10 η ώρα και πρέπει να ψηφίσουμε στις 3 ε, Δεκεμβρίου στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και στις 6 στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Να σας πω ότι βρήκαμε την απάντηση στην ερώτηση που είχαμε θέσει πριν κάποιες εβδομάδες για τον σωστό τρόπο ορισμού των ανθρώπων ε, τουρκικής ε, προέλευσης που ζουν στην Κύπρο. Είναι η τουρκοκυπριακή κοινότητα, έτσι την αναφέρουμε. Αυτό είναι ο ισχύον όρος, ο επίσημος όρος το σχέδιο κανονισμού που μας παρουσίασε και η κυρία Νιέσκη. Ευχαριστούμε κυρία Συγήτρια. Τελευταίο θέμα, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Α, συγγνώμη κυρία Αρτόγκ, είχατε ζητήσει το λόγο για την έκθεση Νιέσκη. Παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ. Χαίρομαι με την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και το σχόλιο της Επιτροπής Ελέγχου γι' αυτό, για την έκθεση της κυρίας Νάινς και μιλώ. Πρόσφατα πήγα στην Κύπρο και ε, είδα διάφορα μέρη και τον ΟΗΕ στην πράσινη γραμμή και το βόρειο τμήμα, το κατεχόμενο και η πράσινη γραμμή καταβάλουν αιτήματα, μάλλον υποβάλλουν αιτήματα ε, σε μας ως βουλευτές να κάνουμε ε, διαβήματα στην Τουρκία για να συνεργαστεί. Είναι ανίποτο πραγματικά αυτό που συμβαίνει. Η Τουρκία να μην συνεργάζεται αυτό τον καιρό λόγω Κυπριακής Προεδρίας με το Κοινοβούλιο και ε, την Κομισιόν. Θέλω να πει η κυρία ε, ότι καταδικάζουμε ε, την τουρκική κατοχή της Κύπρου και το επαναλαμβάνουμε και σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΕ 541 και με δικά μας ψηφίσματα και από το 2006. Επίσης, η χρηματική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλειστικά τώρα θα πρέπει να γίνεται μέσω της νόμιμα αναγνωρισμένης ε, κυβέρνησης που είναι η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι μέσω διαφόρων σκοτεινών ε, και παρανόμων διάβλων στο βόρειο τμήμα της νήσου. Και θα ήθελα να πω ότι αποκλειστικά και μόνο η αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας των ελεύθερων περιοχών ε, θα πρέπει να είναι αρμόδια, θα πρέπει να είναι ο συνομιλητής και εκείνος που φροντίζει να πηγαίνουν ε, σωστά και να γίνεται καλή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ευχαριστώ. Merci. Merci, σας ευχαριστούμε κύριε Χάρτονγκ. Πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Φαντάζομαι θα υποβάλλετε τροπολογίες. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Να καταθέσετε μέχρι αύριο κάποιες τροπολογίες και θα τις εξετάσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί είναι όντως λεπτό το θέμα και πολύ σωστά μας επιθυμήσατε την αδεδηλωμένη θέση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Και πρέπει να ε, εξακριβώνουμε το κατά πόσο οι ενισχύσει που δίνουμε στην ε, τουρκοκυπριακή κοινότητα όντω φτάνουν στον προορισμό τους και δεν είναι ένα έμεσο μέσο ε, αναγνώρισης μίας ε, αρχής που δεν έχουμε επίσημα αναγνωρίσει. Είναι κάτι αντίστοιχο, παρά τις τεράστιες διαφορές κάτι παρεθαρές με το θέμα που είχαμε στην επαλήθευση της βοήθειας προς την Παλαιστινιακή Αρχή. Έλεγχο στο κατά πόσο φτάνει η βοήθεια στους πληθυσμούς που πραγματικά χρειάζονται την αρρωγή μας. Αλλά να μην χρησιμοποιηθεί αυτή η βοήθεια από το άλλο μέρος με το οποίο διαφωνούμε. Περνάμε στο τελευταίο θέμα, τον παραπλησμό των πυρηνικών εργοστασίων σε πολύ σημαντικές χώρες τη Βουλγαρία, πυρηνικό σταθμό του Κοζλοντούι, τη Λιθουανία, η Γκναλίνα. Χθε μάλιστα συνάντησα τον Λιθουανό Υπουργό που μου μίλησε για το θέμα αυτό και ε, τον ποινικό σταθμό της ε, Σλοβακίας, δεν θυμάμαι πώ τον λένε. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που καταφέραμε πριν το, το τέλος της συνεδρίας να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και μάλιστα τόσο 90 λεπτά 35 ε, λεπτά πριν το τέλος της συνεδρίασης. Έχουμε λοιπόν ε, τέτοια πυρηνικά εργοστάσια στη Σλοβακία, Λιθουανία και Βουλγαρία. Είχε συμφωνηθεί ο παροπλισμός τους στις δεξιακές διαπραγματεύσεις των τριών χωρών αυτών και ε, συνοδευόταν από 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ προπολογισμό για τα τρία αυτά σχέδια. Στο μεταξύ απαροπλίστηκαν οι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες και δεν έχουν ενεργοποιηθεί έκτοτε. Παρά τις πιέσεις ε, ε, ε, μετά την κρίση του φυσικού αερίου του 2009, τις πιέσεις από την Ρωσία. Βέβαια υπήρξαν κάποιες ολιγορίες ε, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία παραπλησμού, ιδιαίτερα τη διαχείριση και την τελική αποθήκευση των ε, ε, πυρηνικών αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι 559,2 εκατομμύρια χρειάζονται επιπλέον για να ολοκληρωθεί ο παραπλησμός αυτών των πυρηνικών εργοστασίων με αναλήψει υποχρεώσεων που φτάνουν μέχρι το 2020 και πιστώσεις πληρωμών μέχρι το 2025. Πιστεύουμε ότι είναι δικό μας καθήκον να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν. Α, ναι, Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Και δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στο θέμα αυτό του παραπλήσμου. Το θέμα είναι πόσο καιρό ακόμη και με πόσα ε, κονδύλια θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τέτοιου είδου προγράμματα παροπλισμού. Βέβαια, το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί και από την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Για εύλογου λόγου. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε κάποιε εκτιμήσει ε, για το τελικό κόστος, παρόλο που ε, βλέπουμε ότι μερικές φορές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λάθη. Συμφωνούμε με τα ποσά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που προτιμώ ενδεικτική κατανομή για να έχουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των προγραμμάτων, νομίζω ότι όλοι ε, συμφωνούμε να έχουμε και συγκεκριμένη διορία για το πέρας των προγραμμάτων, να μην το αφήσουμε ανοιχτό αυτό το θέμα του χρονοδιαγράμματος. γιατί και στη Φιλανδία που είχαμε ένα παρόμοιο πρόγραμμα είδαμε ότι έγινε κακή χρησιμοποίηση των κονδυλίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την νομική βάση της χρηματοδότησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ως βάση το άρθρο 203 της Συνθήκης ε, Ευρατόμ με διαδικασία διαβούλευσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τη Λιθουανία ισχύει η ιδιαίτερη βάση, το πρωτόκολλο 4 της ενταξιακής, ε, της ε, συνθήκης, που αποκλεί τελείως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις διαβουλεύσεις. Έχουμε αντιφατικές πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ό,τι αφορά τις συνέπειες του διαχωρισμού ε, των ε, νομικών βάσεων. Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για το πού θα οδηγήσει η διπλή αυτή νομική βάση. Εγώ θεωρώ ότι και τα τρία προγράμματα αρρωγή θα πρέπει να ενταχθούν στην ίδια νομική βάση, να μην έχουμε δύο διαφορετικές, ξεχωριστή για τη Λιθουανία, παρόλο που ε, η αρχική συμφωνία με τις τρεις χώρες ε, είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τώρα, μετά την ε, εξεταστική αποστολή που κάναμε στην Ιγραλίνα, διαπιστώσαμε σοβαρά προγράμματα στη διοργάνωση, παρόλο που το πρόγραμμα ε, παραπλησμού συνεχίζεται. Υπάρχουν ε, και νομικές αντιδικίες για το πρόγραμμα, ειδικά Β1, την, το σταθμό αποθήκευσης των ε, πυρηνικών αποβλήτων. Βέβαια, δεν κάνουμε κάποια γενικά σχόλια, όχι ειδικά για τα συγκεκριμένα προγράμματα, αλλά ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει πίεση στους ενδιαφερόμενους, ώστε να ε, επιληθούν οι νομικές εκκρεμότητες. Ίσως ε, μια λύση θα ήταν να ανασταλεί η χρηματοοικονομική υποστήριξη προκειμένου να ασκηθούν ε, έντονες πιέσεις στις ενδιαφερόμενους είτε να λύσουν την αντιδικία τους είτε να ακυρωθεί το πρόγραμμα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Λιθουανία δεν είναι και πολύ πλουσία χώρα και αν αυξηθεί ο ενεργειακός προϋπολογισμός θα βρεθεί σε ακόμη χειρότερη θέση. Γι' αυτό και προτείνω κάποιες τροπολογίες ε, που περιορίζουν ε, την εμβέλεια της κοινοτική χρηματοδότησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τεχνικές διοικητικές δαπάνες, ε, δαπάνες σε επικοινωνία και πληροφορίες και ούτω καθεξής. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας για ενδεχόμενες απορίες ή και κάποιες ανακριβείς πληροφορίες που ακούμε τις τελευταίες μέρες. Ευχαριστώ κύριε εισηγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, πάρα πολύ συγκεκριμένη η έκθεση αυτή και έχουμε την ευκαιρία να μπορούμε να υποφεληθούμε από την εμπειρία σας και την πραγματογνωμοσύνη σας. Ο κύριος Γκάιερ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν έχω ερωτήσει εγώ στον συνάδελφο Τόρβαλτς μερικές συμπληρωματικέ πληροφορίε από την άποψή μου και ε, από την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών που ασχολήθηκε πάρα πολύ εντατικά με αυτό το θέμα για τα τρία πυρηνικά εργοστάσια. Είναι επίμαχο το θέμα και πολύ. Το πρόβλημά μας ποιο είναι. Μια έκθεση πρωτοβουλίας του κυρίου Μαρινέσκου του ΕΛΚ ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο με μεγάλες αλλαγές, με μεγάλη πλειοψηφία και οδήγησε και αυτό σε έκτακτη έκθεση ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Συναντήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών και συμφώνησε φέτος να μεταβεί στη Λιθουανία και να επιθεωρήσει την Ιγναλίνα και του χρόνου θα πάει και στα δύο άλλα εργοστάσια. Διαλέξαμε πρώτα την Ιγναλίνα, διότι εκεί είναι τα προβλήματα τα, ε, πιο περίπλοκα από τα άλλα μέρη. Επιστρέφοντας από την Ιγναλίνα, διαπιστώσαμε ότι η έκθεση Μαρινέσκου, όπως έχει τώρα, δεν μας βοηθάει πάρα πολύ. Αυτή είναι δική μου άποψη προσωπική. Και είναι επίμαχη η κατάσταση στην Επιτροπή Ελέγχου. Έχουμε μια πολύ στεναρή θέση υπέρ της έκθεσης Μαρινέσκου και μια πολύ στεναρή θέση Λιθουανών συναδέλφων από διάφορες πολιτικές ομάδες που έρχονται αντιμέτωποι και δεν βοηθάει την κατάσταση αυτό όμως για να προχωρήσει η επίλυση του προβλήματος. Υποστηρίζω τις προτάσεις του κυρίου Τόρβαλτς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα. Κάποια στιγμή να τερματιστεί αυτή η κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό έχουμε εμπειρία από τα προγράμματα που μας διδάσκει ότι έχει νόημα αυτοί που καλούνται να παροπλήσουν πυρηνικά εργοστάσια να υφίστανται κάποια χρονική πίεση. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα για την Ιγναλίνα, αλλά εξεπλάγει ως μέλος της αντιπροσωπείας ε, που ε, μίλησα με πέντε συνομιλητές και ο καθένας μου έλεγε διαφορετικό, διαφορετικό υπέτειο για τις καθυστερήσεις. Ε, και ήταν όλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Δεν ήταν μόνο τα συμβαλώμενα μέρη, οι κομισιόν ή και οι κυβερνητικές υπηρεσίες της Λιθουανίας της ίδιας, που μπορεί να είναι και το ελεγκτικό συνέδριο, αν το θεωρήσουμε κυβερνητική, που μας είπαν ο καθένας διαφορετικό λόγο για την καθυστερή κατάσταση. Ναι, εντάξει, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι Το είναι πάρα πολύ περίπλοκα τα προγράμματα. Κανείς ακόμα δεν έχει παροπλήσει ε, ένα τόσο μεγάλο εργοστάσιο και έναν αντιδραστήρα τέτοιου τύπου. Ε, και υπάρχουν και άλλα προβλήματα που οδηγούν σε καθυστερήσεις ολιγορίες, άρα και μεγαλύτερο κόστος. Όλα αυτά είναι κατανοητά και μπορεί κανείς να τα φανταστεί, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε τέρμα. να μην γίνει αυτό το πράγμα ε, συνεχής πληγή που να ζητάει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβάρυνση διαρκής. Θα πρέπει να φαίνεται κάπου το τέλος αυτής της προσπάθειας. Θα ήθελα να ακούσω και τα ποσά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, επίσης να υποστηρίξω τον κύριο Τόλβατ στο θέμα της νομικής βάσης. Εάν σε αυτό το σημείο εμείς δεν ε, έχουμε συναπόφαση στα οικονομικά, υπάρχει κίνδυνος ε, οι εκταμιεύσεις, να το πω προσεκτικά, να ε, διαρκέσουν περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Γι' αυτό ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε να ασκήσουμε πίεση και να έχουμε λόγο για τη ροή των κονδυλίων. Και μπορώ να σας πω ότι είναι απολύτως απαραίτητο και επίγον, γιατί πήγα και εκεί και έχω ήδη άποψη ε, λόγω της αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ. Πραγματικά είναι μαρτυρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα γιατί έχει μεταβεί εκεί επί τόπου. Ο κύριος Ήβαλο Κάλφιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, με την άδειά σας ε, θα μιλήσω υπό διπλή ιδιότητα. Μιλώ και εξ ονόματος της εισηγήτριάς μας που θέλει να εκφράσει τις απόψεις της και πολύ σύντομα ε, θα μιλήσω για ορισμένα από τα θέματα που ανέφεραν ο κύριος Τόρβαντς και ο Γιάννης Κάιερ. Πρώτον, να σας πω τη γνωμοδότηση της Εντίτ Χερσόκ, πολύ σύντομα. Πιστεύει ότι η τελική ευθύνη θα πρέπει να παραμείνει στα κράτη-μέλη, ε, τα αρμόδια για τον παροπλισμό των εγκαταστάσεων. Ταυτόχρονα η οικονομική ευθύνη όμω είναι κοινή μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είχε συμφωνηθεί από την αρχή. Το δεύτερο, πρόβλημα λιγονιών και οι αλλαγές, οι διαρθρωτικέ και οι οργανωτικές πρέπει να λυθούν. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρξει συνολική εκτίμηση ε, και της διαδικασίας της ίδιας του παροπλισμού αλλά και της ε, διαδικασίας ε, μετριασμού και αντιμετώπισης της επίπτωσης που θα έχει το κλείσιμο των εργοστασίων αυτών στην όλη οικονομία της χώρας. Μετά, Υπάρχουν και μια, τεχνικές τροπολογίες που προτείνει για τον προπολογισμό η κυρία Χέρτσοκ. Ε, αφορά και πάλι ενδεικτικά ποσά, όπως είπε ο κύριος Τόρβατς. Αυτό είναι ε, τμήμα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ποσά οριστικά τώρα. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τη δυνατότητα απορρόφησης ε, του εκάστοτε κράτους μέλους. Οι εκταμιεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν κανένα άλλο ενεργειακό πρόγραμμα παρά μόνο τον παροπλισμό πυρηνικών εργοστασίων. Αυτά λέει η κυρία Ντίτερ Χέρτζοκ. Να προσθέσω και εγώ μερικά τώρα σχόλια εξ ονόματός μου για ε, τα θέματα που ακούστηκαν. Βέβαια, τα ποσά θα πρέπει να αποφασιστούν στο PDP, αλλά πρέπει να σας πω ότι τα ποσά αυτά απέχουν πόρο από τις ανάγκες. Να σας δώσω το παράδειγμα με τη χώρα που γνωρίζω εγώ καλύτερα γιατί κατάγομαι από εκεί, μέχρι το 2020 το σχέδιο παροπλισμού θα χρειαστεί 880 εκατομμύρια ευρώ. Η Βουλγαρία ζήτησε τα μισά περίπου, 450 από τον κοινοτικό προπολογισμό. Στην αρχική πρόβλεψη ήταν 208 και τώρα έχουν γίνει 108 από τα 820 που χρειαζόμαστε βάσει του υπολογισμού μέχρι το 2020. Θα πρέπει λοιπόν να τα έχουμε υπόψη μας αυτά. Έχουν κλείσει όλες οι μονάδες πολύ νωρίτερα από ό,τι θα θέλαμε, οπότε ε, δεν έχει συσσωρευτεί ε, πολύ υλικό για να κλείσει. Και επίσης στο Κοσλοντούι δεν υπήρχε καμία τεχνική ε, αιτιολόγηση. Απλώς και μόνο επειδή τότε όταν υπογράψαμε για να μπούμε στην Ένωση δεν ήταν η πυρηνική ενέργεια δημοφιλής ε, στην Ένωση για λόγους πολιτικούς. Και μας ε, υποσχέθηκαν ότι θα καλύψει ο κοινοτικός προπολογισμό το επιπλέον κόστος ή το υπερβολικό. Σε ό,τι αφορά το, το, χρονικό ορίζοντα, την προθεσμία, την καταληκτική και την πίεση τη κυβέρνηση, συμφωνώ. Αλλά υπάρχουν και κάποιε τεχνικέ απαιτήσει. Εγώ δεν είμαι ειδικό στα πυρηνικά εργοστάσια, ούτε στην πυρηνική ενέργεια, αλλά έχω ακούσει ότι υπάρχουν τεχνικοί λόγοι και χρειάζεται μια τεχνολογία να εφαρμοστεί και ε, για τις χρησιμοποιημένες ράβδους και τα κατάλοιπα των καυσίμων. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά έτσι τόσο γρήγορα. Υπάρχουν απαιτήσει ασφαλείας. Το Κοσλοντούι και πάλι σας λέγω θα έχει κλείσει το 2030 οριστικά. Θα έχει τα σχέδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν πούμε λοιπόν ότι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμή θα ήταν το 2020, σημαίνει ότι έχουμε μια δεκαετία τη χώρα στο έρμεο των εξελίξεων να αντιμετωπίσει στο έλεος συγγνώμη, των ε, εξελίξεων ε, ε, και είναι πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση να αντιμετωπιστεί από τη χώρα μόνη της. Και επίσης αυτά που λέει η Edith Herzog αναφέρονται καθυστερήσεις, ολιγορίες, κακοδιαχείριση κτλ. Φοβούμε πάρα πολύ ότι καμιά φορά να μην γνύουμε τις διάφορες περιπτώσεις. Εγώ θα ήθελα να αναφέρουμε, να κατονομάζουμε τις καθυστερήσεις και τις ολιγορίες και να μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Γιατί κάπου μπορεί να υπήρξαν καθυστερήσεις, κάπου όχι. Τα προγράμματα ε, πηγαίνουν καλά, εκταμιεύονται σωστά τα κονδύλια χωρίς προβλήματα ε, και το χρονοδιάγραμμα τηρείται. Δεν είναι όλοι στην ίδια μοίρα. Δεν παίρνουμε το κακό παράδειγμα, ας πούμε, και τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι και για τη νομική βάση. Παρά το γεγονός ότι έχουμε διάφορες πρακτικές σε διάφορες χώρες, συμφωνώ πολύ με τον κύριο Τόρβαλτς, θα πρέπει και εμείς να έχουμε την ίδια νομική βάση και λόγο. Η Λιθουανία κατάφερε να βάλει το θέμα αυτό στη συμφωνία σύνθεσης προσχώρησης μάλλον και θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συμφωνία, τη συνθήκη ε, ερήμην του Κοινοβουλίου. Στις άλλες δύο χώρες υπάρχει ένα χρονικό όριο με ανανέωσή του και συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Αλλά οι τρεις περιπτώσεις είναι αντίστοιχε και εγώ θα συμφωνούσα και με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι μία ενιαία η νομική βάση για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Merci, mon cher collègue. Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κάποια σχόλια. Συμφωνώ με τον βούλγαρο συνάδελφο. Εγώ προέρχομαι από την Σλοβακία και έχουμε μια παρόμοια κατάσταση με την εξαίρεση από ό,τι κατάλαβα όταν έλαβα την επιστολή από τον Πρωθυπουργό μου πριν από κανένα χρόνο ότι η Σλοβακία σίγουρα δεν θα <clears throat> τελειώσει. Το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο 2020. Πιθανότατα δεν θα πάμε μέχρι και το 2030, αλλά και θα χρειαστούμε και άλλα 2-3 χρόνια από το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Σας παρουσίασε την κατάσταση πολύ ξεκάθαρη. Είμαστε σε μια πολύ επισφαλή θέση και οι χώρες είμαστε κάποιες από τις φτωχότερες χώρες της Ένωσης. Δεν θα πρέπει να φεθούμε στη μοίρα μας. Κάτι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό και ελπίζουμε στην αλληλεγγύη από τους συναδέλφους και από τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Βλέπετε κύριε Σιγητά ότι η έκθεσή σας και η παρουσίασή σας έδωσε λαβή για διάφορα σχόλια που μάλιστα συμφωνούν μεταξύ τους. Εγώ προσωπικά να προσθέσω ότι είχα κυβερνητικέ αρμοδιότητε στη Γαλλία όταν αρχίσαμε να διαπραγματευόμαστε με τι άμεσα ενδιαφερόμενε χώρε όσον αφορά τις συνέπειες της τραγωδίας του Τσερνομπίλ για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει τις εν λόγω χώρες συμπεριλαμβανομένες και της Ουκρανίας για να μπορέσουν να κλείσουν αυτούς τους αντιδραστήρες του Τσερνομπίλ που λειτουργούσαν ακόμα, να χρηματοδοτηθεί η σαρκοφάγος που είχε στόχο να εξωτερώσει οριστικώς τον αντιδραστήρα που είχε εκραγεί και να δούμε χώρα προς χώρα και κυρίως αυτές που αναφέρονται τώρα πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε είτε ώστε να εξυγχρονίσουμε στους καλύτερες προδιαγραφές ασφάλειας για τους αντιδραστήρες που ήταν υποκατασκευή και να κλείσουν τελείως οι αντιδραστήρες που δεν μπορούσαν να εξυγχρονιστούν. Και εντυπωσιάστηκα έκτοτε από την μεγάλες προσπάθειες και θυσίες που ζητούσαμε από τις ε, εν λόγω χώρες, γιατί είναι προφανές ότι σε αυτές τις τρεις χώρες, ιδιαίτερα Λιθουανία, Βουλγαρία και Σλοβακία, οι εν λόγω πυρηνικοί σταθμοί προσέφεραν, παρήγαγαν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ηλεκτρισμού που καταναλωνόταν στις χώρες. Μέσα σε λίγα χρόνια χρειάζεται για να κλείσουν και για να προμηθευτούν αυτές οι χώρες ηλεκτρισμό πληρώνουν διπλά τα δαπάνη του παραπλησμού και την αύξηση της τιμής της ενέργειας που οφείλεται στην ε, κατάργηση αυτής της εθνικής παραγωγής. Βασικό καθήκον αλληλεγγύης λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα για τα παλιά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσουν αυτές τις χώρες ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν αυτά τα προγράμματα ανα... μετατροπής ενεργειακής αλλά και της ασφάλισης αυτών των σταθμών που δεν μπορούν να εξυγχρονιστούν. Να προσθέσω, όπως μάλιστα ήδη υπόθηκε, ότι η Λιθουανία θα έχει την ε, Προεδρία το δεύτερο εξάμεινο του επόμενου χρόνου. Μετά από αίτημά του δέχτηκα χθε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ε, του, της Λουθωνίας γιατί ήρθε σε επαφή μαζί μου γιατί είδε πόσες δυσκολίες υπάρχουν για εξέβρεση συμφωνίας για τον ετήσιο προπολογισμό ανάμεσα σε εμά και το Συμβούλιο και αυτό μου επέτρεψε να του εξηγήσω ότι τρέχει, να του πω ότι αν δεν συνεργαστεί και το Συμβούλιο θα βρεθούμε σε δύσκολη κατάσταση για το χρόνο. Όσο μπορούσα τον καθησύχασα για την ε, Λιθουανία και για αυτό το πρόβλημα του παροπλισμού για το οποίο μου μίλησε επί μακρόν, πράγμα το οποίο κατανοώ. Δεν μιλήσαμε για την νομική βάση, αλλά θεωρώ προφανές ότι μια χώρα που σκοπεύει να προεδρεύσει, που πρόκειται να προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμφωνεί στην αρχή μιας δομικής βάσης έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να παίξει πλήρως το ρόλο του. Θα πρέπει να θυμίσουμε τους λόγους για τους οποίους η Λιθουανία αφού ρύθμισε το πρόβλημα όσον αφορά το πρωτόκολλό της ε, αυθορμήτως προτιμά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Αλλά πιστεύω ότι στο πλαίσιο της ε, μεταξύ κυρίων ε, ε, συμφωνίας θα ακολουθήσουμε την πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική λύση. Κύριε Σιγητά, θέλετε να κλείσουμε τη συζήτηση. Uh, Λίγα σύντομα σχόλια. Βρισκόμαστε μεταξύ σφύρας και άκμονος τώρα. Έχουμε, δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τα οριστικά ποσά. Αλλά υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας ή της ανασφάλειας ε, που μας περιέγραψαν ο κύριος ε, Κάλφεν και Στάσνικ ε, σε περίπτωση που δεν ρυθμιστεί το πρόβλημα. Ξέρω τι θα γίνει. Ήμουν δημοσιογράφος και πήγα στο Τσελιαμπίσκ. εκεί είχαμε μια έκρηξη στη δεκαετία του 50 και έγινε πολύ, κακή, πολύ κακός χειρισμός μετά και οι συνέπειε ήταν ε, πολύ αρνητικές. Γνωρίζουμε όλοι πόσο σοβαρά είναι τα θέματα, όχι μόνο από οικονομική άποψη, αλλά και άποψη ασφάλειας. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε οι γαλακτοφόρες για να μας αρμέγουν ε, επαόριστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και η γερμανική παρατήρηση ήταν πολύ σωστή και λογικό είναι να υπάρξει κάποια παράταση αλλά όχι ε, τέρμονο να διονύσετε αυτό το θέμα. Θα ψηφίσουμε στις 28 ε, Νοεμβρίου ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την γνωμοδότησή μας και να ψηφίσει Στη Αρμόδια Επιτροπή Ήτρε 18 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ, από την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ όσους άντεξαν μέχρι το τέλος. Επόμενη συνεδρία 28 Νοεμβρίου, λύεται η Συνεδρία.